Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας με το πρώτο σημείο έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Καθώς δεν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και στη συνέχεια αμέσως μετά έχουμε την έγκριση των πρακτικών από την 6η Δεκεμβρίου, 13 Σεπτεμβρίου, 27-28 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου, 13 Ιανουαρίου, 17 Ιανουαρίου, 24-25 Ιανουαρίου, 1η Φεβρουαρίου και 7η Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχουν εγκρίσεις, κυρώνονται, επικυρώνονται τα πρακτικά. Στη συνέχεια περνάμε στις ανακοινώσεις ε, της Προεδρίας του Πρόεδρου. Λοιπόν, Η σειρά των θεμάτων που θα εξεταστούν σήμερα είναι απόφαση, συνέπεια της απόφασης ε, να επεκταθεί η θεσινή σε σχέση με η ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβουλία στη σημερινή μέρα και σε σχέση με τα κατεπίγοντα καθορισμός, προσδιορισμός ε, μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αναβολή των υπολείπων θεμάτων για τις, 18 ε, τις 18 ε, του μήνα Φεβρουαρίου. Και έχουμε και μία διόρθωση για τον κανονισμό για τις ε, υπηρεσίες αξιολόγησης rating Δευτέρα 14 Μαρτίου αυτό το διορθωτικό το διορθωτικό που υιοθετήθηκε στις 15 σε σχέση με το Κοινοβούλιο διανεμήθηκε σε σχέση με τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Σύμφωνα με τον κανόνα 216 του κανονισμού η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να εξετάσει το σχέδιο με την πρόταση και το διορθωτικό που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να γίνει λόγος για το, την ουσία και τη διαδικασία γιατί είναι γνωστά. Και περνάμε στο σημείο 4 που θα δώσω τον λόγο στη συνέχεια στον κύριο Άκενχόρν που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Συμβουλευτικού Φορέα για την διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ε, θέμα του σειρμού της μόδας στην κρίση που περνάμε. Κυρία Άκερμαν, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, λέει κύριο Άκερχολμ, να παρουσιάσω την ενδιάμεση έκθεση. Είναι η δεύτερη σε μια ολόκληρη σειρά τριών που θα παρουσιάσουμε ως ε, ΕΣΚΑΠ στην αξιολόγηση στατιστικής ε, κατάστασης ε, και διοντολογικού κώδικα και της υλοποίησης του διοντολογικού κώδικα για τα στατιστικά η έκθεσή μας θεμελιώνεται σε αυτά που έγιναν κατά τα παρελθόντα έτη επικεντρωνόμενοι στην ανεξαρτησία, επαγγελματική ανεξαρτησία για την ε, επάρκεια των πόρων και την χρήση, την δέσμευση των κονδυλίων. Σε σχέση με την πρώτη έκθεση προσπαθήσαμε ουσιαστικά να ενδυναμώσουμε τη βάση πληροφοριών μας και το κάναμε αυτό διτά με δύο τρόπους. Αποστήλαμε ερωτηματολόγια στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των χωρών μελών και επίσης προσεγγίσαμε έναν αριθμό εμπλεκόμενων για να έχουμε μια εκ των έξω αξιολόγηση για την δική τους εντύπωση για το ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του κώδικα. Τώρα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ σφόδρα από τα όσα είδαμε. Πρώτα απ' όλα υπήρξε κάποια πρόοδος όμως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Πρωτού πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι υλοποιήθηκε σωστά ο διοντολογικός κώδικας. Δεύτερο, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες NSS ε, ε, δεν θεωρούν πάντα ότι το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στο ύψος ε, των απαιτήσεων, δηλαδή η πρακτική, ας το πω έτσι, καθημερινή εφαρμογή και υπάρχουν ιδιαίτερες επικρίσεις όταν βλέπουν πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Υπήρξε κάποια πρόοδος, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα περίπου 50% των δράσεων βελτίωσης που ταυτοποιήθηκαν έχουν υλοποιηθεί. Αλλά θυμηθείτε ότι αυτό οφείλεται σε μια ολόκληρη σειρά υλοποιήσεις αυτών των κατευθύνσεων. Και έτσι έχουν υποβληθεί μια ολόκληρη σειρά συστάσεων πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Πρώτον, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την τυπική και επίσημη εφαρμογή στην υλοποίηση, που είναι έχει βραδύ ρυθμό σήμερα και πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου η πρακτική εφαρμογή συνάδει με το πνεύμα του κώδικα, όμως από την άλλη πλευρά η νομοθεσία δεν ευθυγραμμίζεται αναγκαστικά με τον κώδικα. Και ίσως πάνω απ' όλα θα πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια η αύξηση της διαφάνειας αληθεύει για τις σχέσεις εργασίας σε σχέση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τις κρατικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία αιτία, ένας λόγος για τον σκεπτικισμό που, με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αυτά τα θέματα. γιατί υπάρχει ανάγκη για μια, ένα τέτοιο συσχετισμό. Αλλά πρέπει να διαφοροποιείται αυτή η ανάγκη σε σχέση με το διοικητικό επίπεδο και το επαγγελματικό επίπεδο. Και αυτό δεν φαίνεται να είναι σαφές ε, σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια που αφορά διορισμούς και απολύσεις σε σχέση με τους γενικούς διευθυντές και ταυτοποιήσαμε, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου υπήρξε μια σύμπτωση μεταξύ αλλαγής γενικού διευθυντή και της αλλαγής κυβέρνησης αυτόματη. Και αυτό θεωρούμε ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο εκ του σύνεγγυς σε μεγαλύτερο βάθος. Επίσης να ενδυναμώσουμε τις, ε, τον ρόλο των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών στις χώρες ως συντονιστών ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των στόχων. Και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε την εισαγωγή εθνικών έσκαψ όπως προβλέπεται από τον κώδικα και όπως έγινε και στην περίπτωση για παράδειγμα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πλευρά των πόρων τώρα έχουμε ήδη μια κατάσταση όπου ένας ολόκληρος αριθμός χωρών αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Αυτό όμως δεν χρειάζεται κανείς να προβλέψει, να είναι ιδιαίτερα ικανός στις προβλέψεις για να δει ότι σοβεί πρόβλημα σε αυτό το πεδίο. Αφενός έχουμε αυξημένη απέτηση, ζήτηση για τη χρήση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, τις αλλαγές κλιματικές, την φτώχεια και πολλά άλλα θέματα. Νέες λοιπόν απαιτήσει στη ζήτηση στατιστικών στοιχείων. Από την άλλη πλευρά Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυξανόμενα προβλήματα με κονδύλια όσον αφορά τους προϋπολογισμούς σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αναμφίβολα θα δημιουργήσει ένα στενό κορσέα, στο πω πολλούς περιορισμούς όσον αφορά το στατιστικό έργο. Τώρα, τούτων λεχθέντων πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στην θέσπιση προτεραιοτήτων. Θα έπρεπε να δώσουμε προσοχή ιδιαίτερα και στην χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλειών. Επίσης θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Και τούτο φυσικά ισχύει και στο εθνικό επίπεδο, αλλά και την εκμετάλλευση δυνατοτήτων που παρέχονται διασυνοριακά παγκόσμια από τις διαφορετικές δραστηριότητες σχετικά. Επίσης να θυμηθούμε, να θυμόμαστε ότι είναι τυπικό ότι οι μελλοντικές αποταμιεύσεις ε, οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις επενδύσεις και αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα θέτει περιορισμούς μακροπρόθεσμα για να υποφεληθούμε δυνατοτήτων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τώρα από την άλλη πλευρά ε, σε σχέση με την ποιότητα φαίνεται ότι λίγα έχουν γίνει. Διερωτόμαστε μήπως υπάρχει απουσία δέσμευσης ε, Βούληση για να γίνει κάτι. Προτείνουμε ότι θα έπρεπε να δημοσιεύονται εναρμονισμένα και απλουστευμένα στοιχεία εκθέσεων σε σχέση με την πτυχή της ποιότητας. Επίσης, οι ποιοτικέ δηλώσεις ή διακηρύξεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό, διότι και αυτό φαίνεται να είναι πάλι κάτι το οποίο υποβάλλεται, υπόκειται σε κάποια αβεβαιότητα όσον αφορά τους εμπλεκόμενους. Δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και στο τέλος τέλος η ποιότητα είναι κοινό στοιχείο. Η εντύπωση που θα αποκομίζει κανείς σε σχέση με την ποιότητα που θα καθορίζει, θα έχει καθοριστική σημασία για την αξιοπιστία και την βασιμότητα των στατιστικών στοιχείων. Για το μέλλον και την τελευταία έκθεση της ομάδας που ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε να συντάξουμε, θα εξετάσουμε περαιτέρω τα ταυτοποιημένα, τα εντοπισμένα προβλήματα και επίσης θα εξετάσουμε του σε μεγαλύτερο βάθος περισσότερο πάλι σε σχέση με τα ερωτηματικά που αναφύονται όσον αφορά κάποιες χώρες πρόσφατα. Επίσης θα αξιολογήσουμε, θα αποτιμήσουμε τα βιώματα τα οποία συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας και θα κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πώς θεωρούμε πώς αντιμετωπίζουμε την από τον ρόλο της, τι μπορεί να κάνει, τι θα, ήταν, θα έπρεπε να κάνει και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα ε, ταυτοποιήσουμε στην τελική μας έκθεση που θα είναι διαθέσιμη το φθινόπωρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά είχα υπόψη να πω εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα μια και ο μιλητής είναι συμπατριώτη μου. Περιμένω για να φορέσετε τα ακουστικά σα. Λοιπόν, θα υπάρξει ερμηνεία, διερμηνεία από τα Σουηδικά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και χαιρόμαστε που θα κάνετε περαιτέρω συστάσεις για την, ε, θα, γιατί θα εκπονηθεί η πολιτική η οποία θα βασιστεί σε αυτές τις συστάσεις. Και πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούν να κάνουν και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συμβάλλουν στην διαδικασία γιατί υπολείπεται τεράστιο έργο για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Έχουμε επίσης ε, μια καλή ευκαιρία για να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να θεσπίσει νέα μέτρα στον τομέα αυτό. Έτσι, οι θύνοντες ε, στη, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θα δεχτούν τις ίδιες πιέσεις, ούτως ώστε να δράσουν. Θα μπορούσατε ίσως ε, να μας ενημερώσετε για τις συζητήσεις που συνεχίζονται στο Συμβούλιο. Ε, και έχω και μία ειδικότερη ερώτηση, επειδή ασχολήσαμε το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης και κατέχεις όλα τα στοιχεία που το συναποτελούν, ήθελα να ε, σχολιάσετε αν γίνεται το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας θα ε, υπάρχουν, θα προβλέπονται και κυρώσεις, πρόστιμα. Ε, πώς ε, θα ρυθμιστεί το πρόβλημα που υπάρχει με το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας μέσα στη νέα μακροοικονομική σκηνή. Θα προβλέπετε κύρωση για τα κράτη-μέλη που παρα χρησιμοποιούν ε, τα στατιστικά στοιχεία ή ε, που προσκομίζουν ε, πλημελή στατιστικά στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά κράτη-μέλη. Επίσης υπάρχει ενιαίος ορισμός για τα παραποιημένα στατιστικά δεδομένα. Τι εστί παραποιημένο δεδομένο θεωρούμε ότι θα πρέπει μέσα στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο να προβλέπεται ένας ορισμός. Εντάξει, δηλαδή θα προβλέπονται κυρίως αν είναι παραποιημένα τα στοιχεία, αλλά ποια είναι αυτά τα παραποιημένα στοιχεία. Και το θέμα είναι αν είναι δυνατόν να ε, προβλεφθεί ε, ένα τέτοιο ε, ενιαίος ορισμός. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτό το συγκεκριμένο ε, ζήτημα. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ορισμό για τις μελλοντικέ εργασίες και για την ε, τυχόν ε, θέσπιση κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ωραία, και εγώ μπορώ να μιλήσω σου ειδικά λοιπόν. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν, αλλά επιτρέψτε μου αφού έχω αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό το τελευταίο θέμα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσει κανείς ποια στοιχεία είναι παραποιημένα, αλλά είναι δύσκολο να αποδείξει κανεί αν εσκεμμένα παραποιήθηκαν τα στοιχεία ή όχι. Άρα για να θεσπίσουμε ένα σύστημα κυρώσεων θα χρειαστεί να συζητούμε εσαΐ σχετικά με το αν ήταν εσκεμμένη, ξαναλέω, ή όχι η παραποίηση των στοιχείων. Από τα στοιχεία που έχουμε, από τις εμπειρίες μας ε, διαπιστώνουμε ότι ε, μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις ε, ένα σετ παραποιημένων στοιχείων, διότι προφανώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν την οικονομική πολιτική και προφανώς θα αποκτούν ε, αυξανόμενη σημασία στο μέλλον τα στατιστικά δεδομένα. Οπότε, όταν προσκομίζονται ε, παραποιημένα στοιχεία καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται ακόμη και η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας ε, και άρα ε, θα δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Τώρα σχετικά με τις κυρώσεις ε, μπορούν να υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις και διοικητικές κυρώσεις αλλά και πάλι εδώ θα συζητούμε παόριστον για να συμφωνήσουμε πώς ακριβώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις αφού πρώτα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα αν ήταν εσκεμμένη παραποίηση ή όχι. θα δούμε ε, αν ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση ε, πώς ακριβώς, ε, αν αποδειχθεί ότι ήταν εσκεμμένη παραπίση, πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο. Τώρα ας περάσουμε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το σύστημα στο σύνολό του έχουμε Αφενός, το θέμα της αξιοπιστίας ε, των ε, στοιχείων που προέρχονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές και αφετέρου τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας σε σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στη Eurostat δηλαδή. Ε, η Eurostat ίδια ε, πρέπει να κάνει κάποιες ε, κινήσεις αλλά δεν μπορεί να φροντίσει ώστε να είναι αξιόπιστα τα στατιστικά στοιχεία που έρχονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές. Υπάρχει βέβαια περιθώριο βελτίωσης σε διάφορους τομείς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Eurostat να επηρεάζει τα όσα συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο. Ε, το θέμα είναι να διαπιστώσουμε σε ποιο μέτρο συνάδουν οι εθνικοί κανόνες ε, περί ε, στατιστικών στοιχείων με τους κανόνες της Eurostat και τους κανόνες που έχουν προβλεφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πάντως προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αλλά ανησυχούμε ε, διότι είναι αργή η υλοποίηση των διατάξεων. Ε, ίσως θα μπορούσε ε, σε αυτό να βοηθήσει το Κοινοβούλιο, δηλαδή να διατηρεί μια πολιτική πίεση μια σταθερή πολιτική πίεση, ούτω ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις σε εθνικό επίπεδο διότι δεν φτάνει να υπάρχουν ε, διατάξεις, νόμοι, πρέπει και να εφαρμοστούν σωστά για να λειτουργήσουν. Σχετικά με το θέμα της οικονομικής ε, διακυβέρνησης που σχολιάσατε, θα δούμε στο μέλλον πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα συλλογής ε, στατιστικών ε, στοιχείων και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο. Το σημαντικό όμως και ήθελα να το τονίσω είναι όπως είδαμε πριν από ένα χρόνο ε, υπάρχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις αν προσκομίζονται ε, κακής ποιότητας ε, στατιστικά στοιχεία. Ε, στην περίπτωση της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη, διαπιστώσαμε ότι το κόστος μπορεί να είναι απίστευτα υψηλό όταν προσκομίζονται στοιχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα και είναι κακής ποιότητας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ήθελα να δραχθώ απλά της ευκαιρία για να αναφέρω τέσσερα θέματα και να δω αν υπάρχει κάποια αντίδραση σε σχέση με εσά για το θέμα της Ελλάδας. Αποκάλυψε, σαν να μην το ξέραμε πιο πριν, μέχρι ποιο σημείο το, σημείο, το θέμα κυρώσεων όσον αφορά την διακυβέρνηση βασίζεται σε αξιόπιστα, πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Για το πακέτο της διακυβέρνησης υπάρχει μια τροπολογία που προβλέπει πρόστιμο για εκείνες τις χώρες που τα στατιστικά του στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα. Και χρησιμοποιώ τον όρο αξιόπιστος εδώ, ε, είτε είναι ε, αυτό εσκεμμένα είτε όχι. Και σε σχέση με τις, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις μου φαίνεται ότι θα αρκούσε να αναφερθούμε στην αντικειμενική ευθύνη σε σχέση περισσότερο με αυτήν παρότι με την κακή λειτουργία των δημόσιων αρχών. Και ένα άλλο θέμα είναι η πολιτική ευθύνη. Για το θέμα της ε, πολιτικής ευθύνης ε, θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει και να ασκεί τον έλεγχο. Αλλά για τις ε, κυρώσεις σε σχέση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι προφανές ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρότι το πρόστιμο, ακόμα και αν εδώ το θέμα της αντικειμενικής ευθύνης απομένει, συμμερίζεστε αυτή τη θέση ή σας φαίνεται μια απόλυτη ή παρεκκλίνουσα ε, τοποθέτηση αυτή. Δεν τα συζητήσαμε αυτά τα θέματα, οπότε η απάντησή μου είναι σε καθαρά προσωπική βάση. Θα επαναλάβω λίγο ίσως αυτά τα οποία έχω ήδη πει μάλλον. Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται ορισμένα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν κάποια πράγματα τα κάνει κανείς πάρα πολύ αυστηρά και ίσως και σχετικά αυτόματα, νομίζω ότι τελικά τα περισσότερα από αυτά εφαρμόζονται με καθαρά πολιτικό τρόπο. Και θα μπορούσα να φανταστώ μία περίπτωση κατά την οποία αυτά τα οποία θα θεωρηθούν εκ των υστέρων παραποιημένα στοιχεία να υπάρξουν ε, χιλιάδες δικαιολογίες τεχνικής φύσεως οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για σαν για τα λάθη του παρελθόντος και για να μην επιβληθούν πρόστιμα. Θα υπάρξουν λοιπόν συζητήσεις, αλλά θα υπάρξουν και ίσως και αποφάσεις, αλλά και πολύ περισσότερες δυσκολίες στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Θα δώσω το λόγο στον Κάρλ και θα ήθελα να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι προτάσεις προετοιμάζει για τα θέματα τα στατιστικά σε σχέση με το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Ίσως είναι ευκολότερο να τα πούμε αγγλικά γιατί η ορολογία αγγλική είναι σχετικά με τα πρόστιμα για την παραποίηση των στατιστικών δεδομένων αυτό που λέω είναι περισσότερο επεξήγηση παρά ερώτηση. Νομίζω ότι στην ουσία εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν άλοφη από ορισμένε κυβερνήσεις. Πολλά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Βέβαια πολλές χώρες μπορεί να παραδεχτούν το συγκεκριμένο θέμα και σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι εφόσον έχει παραδεχθεί μια χώρα ότι έχει υπάρξει πρόβλημα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αν αντιμετωπίσει κανείς μακροπρόθεσμα λίγο τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του πακέτου οικονομική διακυβέρνησης, βασίζεται στην ιδέα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, της αγοράς, της αγοράς ακινήτων και κατά πόσον τέτοια φαινόμενα σε μία χώρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αντίστοιχες καταστάσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει μια σωστή αξιολόγηση και όταν αξιολογεί μια χώρα για να δει αν έχει κάποιο θεωρητικό πρόβλημα επαφίεται και εξαρτάται από την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Απόψή σας λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα είναι ότι ε, υπάρχουν τέτοιου είδους αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ή πιστεύετε ότι οι προσπάθειες που γίνονται ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, δεν τροφοδοτούνται σωστά. Υπάρχουν οικονομικά συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για πολιτικές αποφάσεις. Θα μπορούσα να σχολιάσω σύντομα. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι αν πολλής τα στατιστικά στοιχεία στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι επαρκή έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή αξιολόγηση. Αν δει κανείς το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο δεν έχει σημασία για το αν το ισοσύγιο δηλώνεται σαν 5,5 ή 5,6. Αυτό δεν δίνει κάποια διαφορά. Το θέμα είναι να έχουμε επαρκή στοιχεία για μια σωστότερη κρίση. Το πρόβλημα ακριβώς είναι το θέμα της ποιότητας της συγκεκριμένης αξιολόγησης, της κρίσης την οποία κάνουμε η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη μερικές φορές ή και απαραίτητη. Το πρόβλημα είναι να, είμαστε είναι δεδομένο ότι τα εμπλεκόμενα μέρη κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να δείχνει κανείς μέσω των μακροοικονομικών στοιχείων ότι είναι σε θέση να ελέγξει τις διαδικασίες και είναι σε θέση να εγγυηθεί την ποιότητά τους. Ε, ε, πριν από λίγα χρόνια κάνει μια συνάντηση στις Βρυξέλλες για να θαυμάσουμε τον κελτικό τίγρη και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τι έχουν κάνει τόσο καλά οι Ιρλανδοί ε, για να πετύχουν αυτά που πέτυχαν τότε θα έπρεπε ακριβώς μέσω των μακροοικονομικών ανισορροπιών τις οποίες είχαμε διακρίνει να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους κόδωνες συναγερμού. Δεν το κάναμε. Καλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Η έκθεση της ΕΣΚΑ είναι πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Συμμεριζόμεθα εν πολύ στα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα απλά να προσθέσω κάποιες σκέψεις να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα κείμενο το οποίο θα αντιμετωπίσει κάποια από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν από την Επιτροπή σήμερα το πρωί μεταξύ των οποίων το πώς θα υπάρξει συγκέντρωση και βελτίωση στην συγκέντρωση ποιοτικών στατιστικών στοιχείων σε υψηλά πολιτικά σημαντικά θέματα και έτσι πώς θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε ε, την σωστότερη εφαρμογή του κώδικα αυτού για τα διάφορα κράτη-μέλη και επίσης να δούμε με ποιον τρόπο θα οργανώσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε να ελέγξουμε ακόμα καλύτερα και τα εκ των προτέρων δεδομένα τα οποία προσφέρονται και τα οποία συλλέγονται από τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Εμείς και στα πλαίσια των αλλαγών έχουμε πάρει από το Κοινοβούλιο περισσότερες εξουσίες για έρευνες στις στατιστικές υπηρεσίες και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς θα πετύχουμε μια καλύτερη μορφή ελέγχου των εκ των προτέρων συλλαγωμένων στατιστικών στοιχείων. Ό,τι κατάλαβα μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. μία φορά στα πόδια σου ειδικά. Θα μπορούσα και πάντοτε να μιλάω σου ειδικά, αλλά τέλος πάντων. Ε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η ποιότητα των στατιστικών ε, στοιχείων είναι το θέμα που έθιξε ο κύριος Χάγκλου, αν κατάλαβα καλά. Υπάρχουν ε, λήψεις ε, ποιοτικέ σε κράτη-μέλη που εδώ και πάρα πολύ καιρό διατηρούν, συλλέγουν στατιστικά στοιχεία. Και στη Σουηδία υπάρχει πρόβλημα με τα στατιστικά στοιχεία. Πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να μετρήσει τους διάφορους οικονομικούς δείκτες. Είναι ένα πρόβλημα. πως ε, ε, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η ποιότητα από τις αρμόδιες αρχές ε, και δηλαδή μπορούν να διαπιστωθούν προβλήματα και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ακόμη και ως προς την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Υπάρχει ε, μία πρόταση και την υποστηρίζω να ακολουθήσουμε ε, την ίδια πολιτική όπως ε, στον τομέα του ανταγωνισμού. Δεν χρειάζεται τώρα να κατονομάσω κράτη-μέλη όπου υπάρχει πρόβλημα με τα στατιστικά στοιχεία, αλλά μια καλή λύση θα ήταν να ελέγξουμε αν είναι ακριβή τα στατιστικά στοιχεία και αυτό μπορούν να τα αναλάβουν και οι ίδιες οι στατιστικές αρχές αλλά και τα Υπουργεία Οικονομικών γιατί τελικά αυτοί είναι οι χρήστες των ε, στοιχείων, των στατιστικών στοιχείων. Θέλετε να απαντήσετε. Τελικά δύο ερωτήσεις θέσατε. Ε, η πρώτη σχετίζεται με τις απαιτήσει ε, περί ποιότητας ε, για τα στατιστικά στοιχεία. Κάτα περίπτωση κρίνουμε πώς ακριβώς παράγονται τα στατιστικά στοιχεία και προσπαθούμε να αποτιμήσουμε την ποιότητα. Που προσπαθούμε πάνω απ' όλα να προσδιορίσουμε είναι ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την ποιότητα των στοιχείων και πώς εφαρμόζονται οι διακηρύξεις ποιότητα ε, σε επίπεδο εθνικών κρατών. Θέλουμε στο μέτρο του δυνατού ομοιόμορφα ε, στατιστικά στοιχεία Ε, το 2005 άρχισε να εφαρμόζεται ο νέος ε, κανονισμός ε, και έχουμε υποβάλει μία πρόταση σχετικά με την σωστή υλοποίηση των διατάξεων και των κριτηρίων περί που βλέπονται στον κανονισμό κατόπιν. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα ε, που ανακύπτουν όταν επιδιώκουμε μια υψηλή ποιότητα και εκεί μπορούν να παρέμβουν οι χρήστες ε, όπως είπατε και εσείς των στατιστικών στοιχείων για να ε, αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε ε, για βελτίωση. Γι' αυτό που είπα τον παραλληλισμό με τον τομέα του ανταγωνισμού. Κοιτάξτε, η Eurostat έχει νέες αρμοδιότητες ε, πλέον και σε μια περίπτωση ε, που διαπιστώνει παραβίαση ή μη συμμόρφωση με τον κανονισμό μπορεί να παρέμβει, μπορεί να διερευνήσει την υπόθεση μάλλον να κληθεί να αναθεωρήσει τα ε, στατιστικά στοιχεία που έχει λάβει και ελπίζουμε ότι έτσι ε, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων αφενός και αφετέρου θα ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα να προσκομίζει κάποιος παραποιημένα ε, στατιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. αν δεν έχει ένσταση ε, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των φιλελευθέρων εδώ θα ε, διακόψουμε για λίγο.

Um, uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Έχουμε τέσσερις μέρες με συνεδριάσεις επιτροπών αυτή την εβδομάδα. Τρέχουμε από τη μία επιτροπή στην άλλη. Τώρα έχουμε μία ακρόαση με τον Πίτερ Πράτ για το διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΑΦ αποφασίσε το Συμβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου να συστήσει το διορισμό του Πίτερ Πράτα από την 1η Ιουνίου μια εντολή η οποία θα κρατήσει 8 χρόνια και σύμφωνα με το άρθρο 283 σημείο 2 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΑΦ και εξέδωσαν λοιπόν την θετική τους γνωμοδότηση και η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα αποφασίσει για τον διορισμό του υποψηφίου στη συνάντηση της 24ης Μαρτίου. Τώρα λοιπόν έχουμε μία ακρόαση και η σύστασή μας θα προέλθει ε, από τη δική μας Επιτροπή. Είπαμε στον Πίτερ ότι έχει 15 λεπτά για να κάνει την εισαγωγική του παρέμβαση. Μου είπε ότι ίσως να μην χρειαστεί 15 λεπτά και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Όλοι είδατε το curriculum vitae του Βαν Πράτ. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας εισαγωγικά τώρα. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, είναι μεγάλη τιμή που είμαι ανάμεσά σας σήμερα Συνειδητοποιώ την ευθύνη α, ε, της θέσης ε, η οποία, για την οποία έχω προταθεί. Αν κοιτάξει λίγο κανείς προς τα πίσω στη λειτουργία της Ευρωζώνης, μπορεί να διαπιστώσει ότι έχει λειτουργήσει σχετικά ικανοποιητικά σε σχέση με τον βασικό στόχο, τη σταθερότητα των τιμών. Αν δει κανείς ε, τα σοκ που αντιμετώπισε η Ευρωζώνη, Νομίζω ότι πολλές από τις προσδοκίες που είχαμε για αυτήν επαληθεύθηκαν στα πλαίσια της διαχείρισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια ορισμένες προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επιγόντως. Κάποιες από τις προσκλήσεις αυτές δεν είναι ειδικά για την Ευρωζώνη, προβλήματα στο πιστωτικό σύστημα σαν παράδειγμα που είναι παγκόσμια Κάποια άλλα όμως είναι ε, θέματα ευρωζώνης όπως η ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης. Κάποιες προκλήσεις είναι τεχνολογικής φύσεως, κάποιες άλλες αυστηρά πολιτικές. Και εδώ το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις προκλήσεις οι οποίες αναφέρονται στο θέμα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δεύτερον στη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και τρίτον στα έκτακτα νομισματικά μέτρα που ελήφθησαν από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το πρώτο θέμα λοιπόν, η πρώτη πρόκληση. Είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η σχέση ανάμεσα στη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο την ανάλυση του δεύτερου πυλώνα της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας, ιδιαίτερα τη διάσταση την πιστωτική. Ακούγεται κάτι το τεχνολογικό, πρακτικά όμως είναι πολιτικό γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τον τρόπο εξέλιξης και ανάπτυξης του πιστοτικού κύκλου στις οικονομίες μας. Έχει σημασία να κατανοήσουμε σωστά το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Αυτό είναι κρίσιμο. Ταυτόχρονα όσο αναπτύσσονται τέτοιου είδους μακροοικονομικά μέτρα έχει σημασία να δούμε πώς επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική και πώς καθορίζονται οι ευθύνες στα διάφορα επίπεδα αρχής τα οποία εμπλέκονται. Το δεύτερο θέμα είναι η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Η κρίση έφερε στην επιφάνεια την έλλειψη ε, μια ισχυρή οικονομικής διακυβέρνηση της ζώνης. Γι' αυτό η νομισματική πολιτική έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σαν κεντρικός τραπεζίτης, όχι μόνο σαν Ευρωπαίος πολίτης, αλλά θα ήθελα να σας καλωσορίσω τις πρωτοβουλίες που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για να ενισχύσετε ε, το ε, κομμάτι το οικονομικό το ισχυρό αυτό πλαίσιο, θα έλεγα το ισχυρότερο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης απαιτείται να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν γιατί τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει την εύρυθμη, απόλυτα εύρυθμη λειτουργία της ε, ε, ζώνης και όλες αυτές ε, οι ε, δυσκολίες ήρθαν στην επιφάνεια τη στιγμή, από τη στιγμή κατά την οποία ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση όχι μόνο ε, γιατί το πιστεύω σαν Ευρωπαίος αλλά και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας νομισματικής πολιτικής και θα πρέπει εδώ να προκαλέσουμε την προσοχή και τη συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε όλους τους πολιτικούς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τη σχέση ανάμεσα στην ΕΚΤΑΦ και τις άλλες αρχές, όχι μόνο τις αρχές εποπτείας αλλά και τους Υπουργούς Οικονομικών και τα κοινοβούλια Όλα αυτά θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις επαφές τους. Με τις αλλαγές αυτές της διακυβέρνησης έχει μεγάλη σημασία η ΕΚΤΑΦ να παραμείνει ανεξάρτητη και σε ένα πλαίσιο εντολής σαφέστατα καθορισμένο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των θολών σε εισαγωγικά εντολών που έχουν δοθεί στις διάφορες αρχές εποπτείας. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνονται οι επαφές ανάμεσα στις διάφορες αρχές και τα επίπεδα αρχής, αλλά να ξεκαθαρίσουμε πριν γίνει αυτό τις βασικές αρμοδιότητες της κάθε αρχής. Η τρίτη πρόκληση είναι η εξομάλυνση των νομισματικών πολιτικών. Όπως ξέρετε η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συνέλθει από την βαθύτατη χρηματοπιστωτική κρίση την οποία αντιμετώπισε και οδηγήθηκαν τα επιτόκια σε πάρα πολύ ε, χαμηλά επίπεδα που δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Θα πάψουν να ισχύουν ε, μέτρα τα οποία ήταν ιδιαίτερα έκτακτα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστός χρονισμός για όλα αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για τις αρχές, ιδιαίτερα στο πάρον πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και επίπεδα, θα έλεγα, ιδιαίτερα ευάλωτα οι προκλήσεις της ΕΚΤ είναι δύσκολες και πολλές, αλλά η συλλογική λειτουργία της και η επαγγελματικότητα των στελεχών της την βοηθούν ιδιαίτερα. Η ΕΚΤ και το διοικητικό της συμβούλιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσικά και την εμπειρογνωμοσύνη και επαϊοσύνη των κεντρικών τραπεζών των ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό είναι σημαντικό οπλοστάσιο. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, εγώ μπορώ να τα αντιμετωπίσω, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και σε πιστοτικό επίπεδο και σε επίπεδο δημοσιοπαλληλικό και σε επίπεδο τραπεζικό και σαν οικονομολόγος στο Δέλτα Νιτάφ ήμουν, καθηγητής οικονομίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και δίδαξα την οικονομία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την επιχειρηματική ιδεοντολογία. Δούλεψα επίσης σε πάρα πολλές μεγάλες βελγικές τράπεζες και αυτό μου έδειξε ακριβώς τις διαστάσεις που έχει το πιστοτικό σύστημα και επίσης ο πολιτισμός ο πιστοτικός θα έλεγα. Από το 1999 με το 2000 ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών και το 2000 πήγα στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου σαν εκτελεστικός διευθυντής υπεύθυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον έλεγχο των συστημάτων πληρωμών. Είμαι επίσης μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Βελγικής Εποπτείας Επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ε, ασχολούμε στα πλαίσια της κεντρικής τράπεζας με την ασφάλεια ε, ε, με την εγγύηση μάλλον των ασφαλιστικών θεμάτων και προσπαθούμε με τους λίγους πόρους που έχουμε να ελέγξουμε και να ορίσουμε τη σωστή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία δέκα χρόνια ήμουνα μέλος επίσης σε πάρα πολλά υψηλά, υψηλού επίπεδου σώματα οικονομικά στην Ευρώπη ε, σε επίπεδο ρυθμιστικό. Απέκτησα θα έλεγα ε, υψηλά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνη σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας, ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων πληρωμών και κατανοώ νομίζω αρκετές επαγγελματικές διαφορετικές νοοτροπίες και σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών και σε επίπεδο ιδιωτικών τραπεζών και σε επίπεδο κυβερνητικών στελεχών. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για να δώσω απαντήσεις. Συντώ συγγνώμη από τη διερμηνία, θα προσπαθήσω να μιλώ πιο αργά στις απαντήσεις μου. Δημιουργήσατε κάποιο πρόβλημα στους διερμηνείς. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις εδώ μπροστά μας. Πρώτη ερώτηση, ε, ο Ζαν Πολ, ε, σε αυτό το γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Άκουσα όλες τις τεχνικές ε, διευκρινήσεις και θέλω να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Πρέτη. Για ποιο λόγο ε, δηλώσατε υποψηφιότητα για αυτό το αξίωμα. Απάντηση. Δύσκολο το ερώτημά σας, όντως διότι σχετίζεται με την ίδια μου την ιδιοσυγκρασία. Είναι πολύ προσωπικό το ζήτημα. Ε, Μπορώ να σας πω ότι όταν οι υπουργοί στο ΕΚΟΦΗΝ ε, με, μου πρότειναν, με πρότειναν για αυτή τη θέση, με ομοφωνία σχεδόν, με πήραν τηλέφωνα οι φίλοι μου και μου είπαν έλα να το γιορτάσουμε. Ε, αλλά εγώ το, τι τους απάντησα, ότι δεν έχει περατωθεί η διαδικασία πρώτον και δεύτερον, όλα ε, αυτά τα συναισθήματα που ένιωθα, ε, ουσιαστικά μεταφράζονται σε ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης ε, για το αξίωμα αυτό ένα από τα ιδανικά μου είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εν πάση περιπτώσει αυτό που νιώθω δεν είναι αν πάμε να γιορτάσουμε, είναι ότι θέλω να επομιστώ πλήρως ε, τις ευθύνες μου. Βλέπετε λοιπόν πώς αντιμετωπίζω αυτή τη θέση. Κοιτάξτε, να προσθέσω ότι γνωρίζω πολύ καλά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ και 10 χρόνια ε, πηγαίνω και έρχομαι στην ΕΚΤ, οπότε ε, είναι μια λογική συνέχεια. Βρίσκω να αναλάβω αυτή τη θέση, αλλά πάντως ε, αυτό που με διακατέχει είναι ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης σε σχέση με τα ε, καθήκοντα. Ε, αλλά ήταν δύσκολο το ερώτημά σας. Ε, ευχαριστώ. Ούγκο. Ούντο. Ούντο Μπούλμαν, ευχαριστώ πολύ Σάραν. Κύριε Πράτ, έχουμε μια νέα κατάσταση από την προηγούμενη εβδομάδα. Από τότε που τα ευρωκράτη συμφώνησαν σε ένα μόνιμο σταθεροποιητικό μηχανισμό που θα εισαχθεί που θα ενδυναμώσει το ευρώ, θα αποτρέψει κρίσεις στο μέλλον. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε στην εισαγωγή σας γι' αυτό, το ότι η νομισματική πολιτική αντιμετώπιζε υπερβολικές προκλήσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπιζε υπερβολικές προκλήσεις γιατί η πολιτική της είχαν, την είχαν εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε ένα σταθεροποιητικό μηχανισμό που θα επέτρεπε στην, στην πρωτογενή αγορά για, για το χρέος να δραστηριοποιηθεί. Με ενδιαφέρει ποια είναι η άποψή σας για τον επιμερισμό έργου μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτού του νέου ESM ε μηχανισμού, δηλαδή νέου μηχανισμού που θέλουμε να δημιουργήσουμε ώστε το ευρώ μακροπρόθεσμα να σταθεροποιηθεί. Ποιο θα αναλάβει ποιο ρόλο ω έργο στον επιμερισμό και πώ οι δύο αυτοί θα συντονίζονται. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Οι συζητήσει φυσικά δεν έχουν ολοκληρωθεί καθοριστικά, τελεσίδικα. Θα απαντήσω υπό το πρίσμα των όσων γνωρίζω και διαισθάνομαι. Είναι σαφές όπως επαναλάβατε ότι η νομισματική πολιτική είχε υπερβολικά υποστεί φόρτο εργασίας και για την ανάπτυξη του νέου μηχανισμού που θα ε, δώσει την δυνατότητα στις κεντρικές τράπεζες να επικεντρωθούν στον αρχικό τους ρόλο, την νομισματική σταθερότητα. Αυτό είναι το κύριο θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Αυτό εξηγεί φυσικά γιατί η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο πρόεδρος της εξέφρασαν την άποψη ότι η ελαστικότητα όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα πρέπει να είναι στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσκαλούσαμε. Θα εκκαλείτο το νέο ESM να ασκήσει εξουσία, αλλά θα πρέπει να έχει επαρκή ελαστικότητα στη λειτουργία του αυτός ο μηχανισμός. Βλέπουμε σαφώς ε, το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός, να μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά χρέους ε, διαφορετικών χωρών στο πρόγραμμα όσον αφορά τα, ε, τα ασφαλιστικά. Είναι ένας ε, προσωρινός μηχανισμός και η διέξοδος ε, από αυτά τα μη ορθόδοξα μέτρα θα πρέπει να διαφαίνεται και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συζήτηση σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και την Υπουργού Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει κέρια σημασία να ολοκληρωθούν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα το μήνυμα το οποίο αποστέλλεται είναι ότι το ESM θα πρέπει σχετικά να έχει ένα ευρύ πεδίο μέσων και δράσεων για να λειτουργήσει σωστά. Αν δεν συμβαίνει αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πούμε ότι θα ε, αντιμετωπίζει υπερβολικές προκλήσεις αν δεν μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν σωστά. Το άλλο σημείο το οποίο αναφέρατε είναι, θα έλεγα, το ότι όταν τα βλέπει κανείς από τα από το εσωτερικό. Είναι δύσκολο να εξευρεθεί η σωστή αλληλεγγύη, για την, η σωστή ισορροπία για την αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουμε στην Ευρωζώνη. Αλλά πρέπει τα κίνητρα να είναι τα ορθά και να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και υπευθυνότητα. Και είναι η όλη συζήτηση. Πού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ των δύο. Πώ μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ουσιαστικά μια πολιτική ήσυφή συζήτηση. Το να βρούμε τα σωστά κίνητρα, τη σωστή ισορροπία μεταξύ κινήτρων και αλληλεγγύη, είναι ένα κέριο ε, σημείο και εσείς θα διαδραματίσετε κύριο ρόλο σε αυτό. Και θέλω να επαναλάβω μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε, όταν επικεντρωνόμαστε σε όλη αυτή τη πολιτική συζήτηση, στο τέλος τέλος απορρέει κάτι που είπα στη σύντομη εισαγωγή μου. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει επαρκής, ας το πω έτσι, απήχηση στους Ευρωπαίους πολίτες και την εμπλοκή τους. Να μην έχουμε μία εκ των άνω προς τα κάτω επιβολή κανόνων ε, για όσον αφορά αυτά τα θέματα αλλά εκ των κάτω προ τα άνω να μπορούν να εμπλέκονται επαρκώς ε, οι πολίτε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ διαδραματίζει ρόλο κλειδιού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που ε, ήθελα να δώσω. Είναι και ένα κύριο σημείο και για την ΕΚΤ διότι ο στόχο τη είναι η νομισματική η σταθερότητα και όσον αφορά τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή τη, λόγω τη νομισματική κρίση, πιέστηκαν τα πράγματα και είδαμε τώρα εδώ ανορθόδοξα μέτρα νομισματικής πολιτικής ε, όσον αφορά την ε, δράση. Ευχαριστώ. Right, thank The question Σας ευχαριστώ από τους φιλελευθέρους. Ε, ποιος θα κάνει την πρώτη ερώτηση, Σιλβή, παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Πράτε, εδώ είμαι. Σωστά επιμείνατε στην παρέμβασή σας στο στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πώς την αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Για να διατηρηθεί ανεξαρτησία της ε, πρέπει και εδώ κάνω μία παρένθεση, γιατί έχουμε συζητήσει με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε ακροάσεις που έγιναν. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ε, καλύψουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον ουσιαστικό πληθωρισμό και την ε, ευρύτερη εντύπωση που έχουμε για τον πληθωρισμό, για τον ποσοστό πληθωρισμού. θα μπορούσατε ίσως να βελτιώσετε τους δείκτες. Ε, δεν είναι ε, καθαρά τεχνικό το ζήτημα, αλλά υπάρχουν και κάποια τεχνικά στοιχεία που πρέπει να δώσετε στην απάντησή σας. Απάντηση. Όταν κάνετε μια ε, δημοσκόπηση σχετικά με τις ε, προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι μάλλον ε, καθησυχαστικές οι απαντήσεις, οπότε δεν έχω την ίδια εντύπωση με σας. Βέβαια, Εάν πηγαίνετε εσείς και ε, κάνετε αυτή την ερώτηση στα, στις διάφορες χώρες, ε, παίρνετε ανάμεικτες απαντήσεις. Σε παράδειγμα, χάρη, ρωτάτε τι πιστεύετε για την αύξηση των τιμών. Ε, έχουμε συστηματικά ένα βαρόμετρο που δείχνει ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικά τα σημεία. Αυτό δεν συνάδει βέβαια με την εντύπωση που έχουμε όταν συζητάμε με του ανθρώπου σε καθημερινό επίπεδο. Πώ μπορώ να απαντήσω. Υπάρχει συχνά μια σύγχυση ανάμεσα στην έννοια τη αγοραστική δύναμη, δηλαδή με το μισθό που έχω, με την αμοιβή που έχω, ποιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών ε, μπορώ να αποκτήσω. Και υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα ε, στην εντύπωση που έχουμε για την αύξηση των τιμών και εκεί είναι μάλλον καθυσυχαστικές οι απαντήσεις ε, ε, και από την άλλη πλευρά έχουμε το πραγματικό μισθό, την πραγματική αγοραστική δύναμη τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ε, οξύνονται οι ανισότητες ε, ως προς τις μισθολογικές, ε, εισοδηματικέ μάλλον διαφορές και έτσι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει την εντύπωση ότι δεν σημαίνεται αύξηση στην αγοραστική παρότι δεν υπάρχει μεγάλη διακύμανση τιμών. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην αγοραστική δύναμη, στον πραγματικό μισθό μου και την γενικευμένη εντύπωση σχετικά με τις τιμές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε να δει αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στους δείκτες των τιμών σε σχέση με το καλάθι του καταναλωτή δηλαδή και είδαμε από τους δείκτες ε, των τιμών ε, μικρές ε, διαφορές χρησιμοποιώντας αυτόν τον δείκτη, το ξαναλέω. Ε, βέβαια πρέπει να επικαιροποιούμε διαρκώς τις μελέτες γιατί στα, στα χαμηλά εισοδήματα φυσικά τα τρόφιμα παραδείγματος χάρη έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο καλάθι των αγαθών σε σχέση με άλλες πληθυσμιακές τάξεις και μπορώ να καταλάβω ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχουμε την εντύπωση ότι έχει, έχουν αυξηθεί οι τιμές περισσότερο από ό,τι μας δείχνει ο δείκτης για το σύνολο του, του, του πληθυσμού. Ε, ίσως θα έπρεπε να κοινοποιούμε, να δημοσιεύουμε ε, σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφορίες που συλλέγουμε στην τράπεζα. Ε, τώρα η ΚΕΙΤ από πλευρά των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Να σας καλωσορίσω λοιπόν με τη νέα σας ιδιότητα. Ευχαριστώ για τις προηγούμενες προηγούμενες φορές που μας έχετε βοηθήσει έχουμε κατανοήσει καλύτερα προβλήματα ε, χρηματοπιστωτικά με τη δική σας σύνδρομη. Εκπρόσωποι της τράπεζας πρόσφατα είχαν έρθει να συζητήσουν μαζί μας από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας την άποψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τα θέματα της ρευτότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι και αυτό μια ευθύνη και ποια ακριβώς θα είναι ε, η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τον έλεγχο ο οποίος θα γίνεται ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και τι ρόλο θα κληθεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν παροχέας θα έλεγα σε εισαγωγικά ρευστότητας προς τα πιστοτικά ιδρύματα ή θα οδηγήσει σε μια αλλαγή ίσως και την κατάργηση των ενδιαμέσων μηχανισμών. Όπως γνωρίζετε μπλέκομαι στις συζητήσεις μέσω της Επιτροπής της Βασιλείας και στην Ευρώπη έχουμε μια επιτροπή ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες, την PSC το Σαββατοκύριακο είχαμε συζητήσει το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε και οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να πω το εξής. Είδατε στο, στο curriculum μου είμαι υπεύθυνο διατάκτης θα έλεγα για θέματα πληρωμών όχι για ανταλλαγές αλλά για τα λεγόμενα clearing στον τομέα της Κεντρικής Τράπεζας λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να υπάρχει σωστή λειτουργία των, δημοσιο... των ε, χρηματοπιστωτικών υποδομών. Είναι δική μας ευθύνη αυτό. Λέμε λοιπόν ότι θέλουμε να εμπλακούμε και στην σύνταξη των επιπέδων τα οποία θα πρέπει να αφορούν όλες τις πληρωμές, τα clearing και τα συστήματα α, α, ρύθμισης του συμψηφισμού Έχουμε εμπλακεί και σε διεθνείς επιτροπές όπως ε, το CPSS. Θέλουμε να συνεχίσουμε την εμπλοκή μας αυτή. Είπα στη σύντομη εισαγωγή μου ότι γνωρίζω εντελώς διαφορετικές επιχειρηματικές αντιλήψεις. Ίσως το έχετε δει και εσείς αυτό όταν βλέπετε οι κεντρικοί τραπεζίτες να ασχολούνται με το θέμα της εποπτείας των υποδομών είναι μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τον έλεγχο οι ελεκτές από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο πολιτισμός, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα είδος στρατιωτικού πολιτισμού, στρατιωτικής κουλτούρας που ε, είναι μία μορφή επίβλεψης χωρίς καμία διακοπή και αυτό προέρχεται από την κουλτούρα των πληρωμών την οποία έχουμε γιατί είμαστε βασικοί υπεύθυνοι σε σχέση με την σωστή λειτουργία του συστήματος πληρωμών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν το θέμα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υποδομών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα πλαίσια της υποδομής που αφορά τα CCP. Το δεύτερο θέμα αφορά την παροχή ρευστότητα. Ξέρετε ποιε είναι οι συζητήσει. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία λέγει ότι τα CCP ε, μπορεί να χρειάζονται ρευστότητα, ε, ενέσει ρευστότητα σε έκτακτες ε, συνθήκες. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Αλλά σε ποιο στάδιο μπορεί κανείς να να διασφαλίσει το πότε θα χρειαστούν τη συγκεκριμένη ρευστότητα. Θέλουμε ακριβώς τα CCP να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε επίπεδο ρευστότητας και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι αν τυχόν όποτε έχετε προβλήματα ρευστότητας θα σας τα παρέχουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν λειτουργεί έτσι. Προσπαθούμε εμείς να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί έτσι ώστε τα CCPs να μην, να μην αντιμετωπιστούν σαν τράπεζες, σαν πιστοτικά ιδρύματα απλά. Κάποιοι από τους συνάδελφούς μου πιστεύουν ότι θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα και με πιο συγκεκριμένο ε, τρόπο το καθεστώς των τραπεζών, περιορισμένο στόχο, Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο και απλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η παροχή ρευστότητα κάτω από συνθήκες πίεσης μπορεί να παρέχεται και πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο, το λειτουργικό έτσι ώστε κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Αλλά δεν θα πρέπει τα CCP να αντιμετωπίζονται σαν πιστοτικά ιδρύματα. Όλοι πάντω συμφωνούν ότι κάτω από συνθήκε πίεση, τα CCP μπορεί να απαιτούν ρευστότητα. Το θέμα είναι αν κάτι τέτοιο θα είναι κάτι το συνηθισμένο, είναι κάτι για το οποίο θα υπάρχουν εκ των προτέρων ρυθμίσεις. Ε, είναι ένα θέμα δύσκολο και γίνεται μια ευαίσθητη συζήτηση για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τα CCPs. Κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι ένα τέτοιο ίδρυμα που ασχολείται με ευρώ θα πρέπει να έχει έδρα στην χώρα ή στην ζώνη στην οποία η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να παρέχει την ρευστότητα που απαιτείται κάθε φορά. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι τέτοια θέματα μπορεί να ρυθμιστούν μέσω των ρυθμίσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν ένα CCP λειτουργεί στο Λονδίνο και λειτουργεί με euro, μπορεί να γίνει με swaps ανάμεσα στις διάφορες κεντρικές τράπεζες. Λοιπόν, δεν θα σας πω ποια θα είναι η κατάληξη στη συζήτηση αυτή, γιατί δεν την έχω ακόμα. Το τελευταίο σημείο. Είχατε και μια τρίτη ερώτηση. Αφορά τη σχέση ανάμεσα στην ΕΣΜΑ και τις κεντρικές τράπεζες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει στενή σχέση ανάμεσα σε αυτές. Νομίζω ότι οι υποδομές είναι είτε ευρωπαϊκές είτε διεθνείς. Σας είπα ήδη από πριν ότι πιστεύω ότι οι δύο αυτές αρχές θα πρέπει να εμπλακούν και οι δύο και θα πρέπει να συνεργάζονται ε, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να διαβουλεύονται απλά, αλλά θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο ε, για το αν θα πρέπει να δοθεί περισσότερη αρμοδιότητα στην ΕΣΜΑ η οποία παίζει ένα βασικό ρόλο. Τελικά αν κάτι δεν πάει καλά σε ένα CCP η Εθνική Αρχή είναι αυτή η οποία έχει την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όλα αυτά είναι λοιπόν θέματα περίπλοκα, δεν μπορώ μέσα σε δύο λεπτά να δώσω απαντήσεις στα θέματα αυτά. Αναγνωρίζουμε πάντως ότι στον τομέα αυτό η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει αρκετές αρμοδιότητες μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου οι εθνικές αρχές να εμπλόκονται και αυτές, γιατί κάποιοι θα πρέπει να λάβουν την πρωταρχική ευθύνη σε περίπτωση κρίσης και εδώ εμπλέκονται και οι κεντρικές τράπεζες οι οποίες θα παρέχουν τη ρευστότητα προς τα CCP κάτω από συνθήκες κρίσης. Λοιπόν, η ανησυχία μου εδώ είναι ότι οι προθεσμίες που έχουμε βάλει ε, το τέλος του 2012 του 2012, λέει το 2002 κατά λάθο ο μιλητής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για διάφορους λόγους και τους λόγους τους οποίους σας εξέθεσα πριν. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εδώ. Τι θα εντάξει κανείς στα CCP στο θέμα των επιπέδων, των κοινών επιπέδων, της ε, αξιοποίησης, του χαρακτηρισμού των διαφόρων επιπέδων CCP από τα κράτη-μέλη κτλ. Θέλουμε και εσείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσετε έτσι ώστε να αλλάξει το τοπίο και να περάσουμε κάπως σε πιο συγκεντρωτικές ε, εμπλεκόμενες πλευρές ε, ε, για να βελτιωθεί ο έλεγχος. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, είναι μια πραγματική πρόκληση. Ήταν πολύ περιπλοκή ερώτηση και καλά κάνατε και μακρηγορήσατε στην απάντηση. Δεν βλέπω κανέναν από τους πράσινους. Γκουε. Ούτε. Godfrey Μπλουμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πράτ. Στην αρχή είχαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Είχαμε τα κριτήρια, τα νομισματικά για όσους προσχωρούσαν ή ήταν να προσχωρήσουν. Και τώρα έχουμε επαναγορά δημοσίου χρέους στη δευτερογενή αγορά. Ε, δηλαδή υπόθηκο δημόσιο χρέος. Με αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα της συνθήκης ε, του Μάστριχτ. Παρόλα αυτά, θεωρείται η συνθήκη αυτή ως ε, εντολή που επιτρέπει δράση ε, για τις ε, κυβερνήσεις. Γιατί αυτές θα χρηματοδοτήσουν τους άλλους τα όσα προβλέπονται. Δεν βλέπετε ότι έχει αποτύχει αυτό το νομισματικό πείραμα. Ούτως ή άλλως ήταν μοιραίο. Ποιο είναι το εφεδρικό σα σχέδιο, αν έχετε εφεδρικό σχέδιο. Απάντηση να σας πω κάτι για τα μη συμβατικά μέτρα που έχουν λάβει, αναλάβει όλες οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δείτε τα στοιχεία θα διαπιστώσετε ότι οι ισολογισμοί κάποιων κεντρικών τραπεζών έχουν σημειο σημαντικότατη αύξηση και αν δείτε το ενεργητικό ε, στους ισολογισμούς, Ας δούμε τη ΣΥΠΑ παραδείγματος χάρη. Θα δείτε μαζικές επαναγορές χρέους στη δευτερογενή αγορά συνήθως διαρθρωμένων προϊόντων που σχετίζονται με τη ακίνητα. Ε, ξέρω ότι ρωτήσατε για την Ευρωζώνη. Ήθελα να θέσω το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης κάποιες κεντρικές τράπεζες και ευτυχώ όχι ευρωπαϊκοί διάφορες κεντρικές τράπεζες ήταν βασικοί αγοραστές στη δευτερογενή αγορά για κινητές αξίες που βασίζονται σε ακίνητα. Ε, και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η αξία αυτών των προϊόντων. Είναι σαφές τώρα, όπως είπατε και εσείς, ότι για ένα, ε, αυτό ισχύει για ένα μικρό κομμάτι του ισολογισμού ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, διότι η αύξηση παρατηρείται στην ΕΚΤ σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά με τι εγγυήσεις, τα collaterals δεν είναι το ίδιο με την Τράπεζα της Αγγλίας, δεν είναι το ίδιο που κάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον ΗΠΑ, αν κάνετε τον παραλληλισμό. Ε, οπότε ε, χαίρομαι για την τάση που παρατηρείτε στην Ευρωζώνη. Τώρα αυτό το μικρό κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, κοιτάξτε, ε, ο στόχος μέσα σε μια ζώνη ενίας νομισματικής πολιτικής ήταν να έχετε το μηχανισμό μετάδοσης, έτσι τον ονομάζαμε, δηλαδή όταν ορίζετε την ισοτιμία πρέπει να δείτε πώς όλες, όλα τα νομίσματα θα ενταχθούν μέσα στο σύστημα και για κάποιες χώρες δεν λειτουργήσε αυτός ο μεταβατικός μηχανισμός ε, εξού και η προσωρινή ε, επέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και ξέρω πώς λένε το συνάδελφο στον Νούντο όταν απαντούσα λοιπόν το είπα αυτό ναι. αυτό έχει κεντρική σημασία για την ΕΚΤΕ, δηλαδή να αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας και δείτε και τις ε, ε, τα διαρθρωτικά εθνικά προγράμματα σε κάποιες χώρες πώς σχετίζονται με αυτό. Ε, φυσικά ελοχεύουν κίνδυνοι για τους ισολογισμούς δηλαδή, αλλά είναι μετρημένοι, είναι υποέλεγχο αυτή η κίνδυνη και είπαμε σε σχέση με τα όσα συζητούνται ε, στο ΕΚΟΦΗΝ ε, ότι συνδέονται άμεσα με την δική σας ερώτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα και εγγεγραμμένος. Τώρα εσείς ε, κύριε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φρέτε. Έχετε μακρά πείρα στην Βελγική Εθνική Τράπεζα και ανεβαίνετε μια βαθμίδα ανώτερα. Και για τις αγορές ομολόγων χρεογράφων αναφερθήκατε ήδη. Έχω ένα άλλο ερώτημα. Πώς κρίνεται το θέμα της νομισματικής σταθερότητας αντιμετώπισης του πληθωρισμού με άλλους στόχους, πλήρη απασχόληση, ε, πρόθεση της ζήτησης, ε, ε, συγκυριακή υποστήριξη οικονομική. Πώς βλέπετε αυτά τα θέματα σε σχέση με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και πώς κρίνεται το σύμφωνο για την σταθερότητα του ευρώ, την ανταγωνιστικότητα του ευρώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτο ερώτημα. Θα έκπιζα, θα σκεφτόμουν ότι θα πηγαίνατε όχι στο παραδοσιακό ερώτημα σε σχέση με την καταπολέμηση του πληθωρισμού και των άλλων στόχων, δηλαδή απασχόληση και ανάπτυξη που είναι η ερώτησή σα τώρα. Σκεφτόμουν ότι η πιο δύσκολη συζήτηση σήμερα θα ήταν η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και η νομισματική σταθερότητα, μια νέα διάσταση τη νομισματική πολιτική. Να δούμε σε ποιο βαθμό επαρκεί η νομισματική σταθερότητα όταν βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ του κύκλου ε, δράσεων του τζίρου επιχειρήσεων και των οικονομικών κύκλων που οι οικονομικοί κύκλοι μπορεί να έχουν μεγάλη, διάρκεια. Δεν σκέπτομαι ότι υπό τους όρους ε, νομισματικής σταθερότητας δηλαδή για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης υπάρχουν πολλά να πει κανεί. Έχει κύρια σημασία ο στόχος νομισματικής σταθερότητας, ε, ο στόχος της συνθήκης να επιτευχθεί. Το βλέπουμε αυτό με σαφήνεια σήμερα, ότι όταν είναι σταθερές ε, οι προσδοκίες όσον αφορά την εξέλιξη του πληθωρισμού, παρέχεται μεγάλο περιθώριο δράσης στην Κεντρική Τράπεζα. Να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα για να υποστηρίζεται ο κύκλος ο επιχειρησιακός. Όμως με όρο και προϋπόθεση την επίτευξη του πρώτου στόχου. Φανταστείτε και όχι μόνο στην Ευρωζώνη αυτή τη φορά αλλά και σε άλλα επίπεδα την κατάσταση που θα δημιουργείται αν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ήταν υψηλότερες όπου οι κεντρικές τράπεζες θα χρησιμοποιούσαν μη ορθόδοξα μέσα, μη συμβατικά μέσα. <clears throat> Και ξέρουμε ότι έχει πολλά να ε, επομιστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε σχέση και με το συμβατικό της ρόλο. Υπάρχουν όρια για το τι μπορεί κανείς να κάνει. Υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν περνάει κανείς σε μη συμβατικές πολιτικές, διότι τα γεγονότα θα το απαιτούσαν αυτό. Η αξιοπιστία όλη τη νομισματική πολιτική να κατοχυρώνεται από πλευρά ε, τη υποστήριξη των πολιτών με, την αξιοπιστία του. Και σε σχέση με το θέμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώ αντιμετωπίζουν τι προσδοκίε πληθωριστικέ προς, προς, ε, οι πολίτε και το πουβουάντα σά, την αγοραστική δύναμη και τι αισθάνονται οι πολίτε. Γι' αυτό όταν βλέπουμε την εξέλιξη των μισθολογικών εξελίξεων, τη ε, πληθωριστική εξέλιξη, συνειδητοποιούμε και τη συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία και τι διαπραγματεύσει που συνεπάγεται αυτό. Αυτό συνδυάζεται με την νομισματική σταθερότητα. Δεν είναι τίποτα το καινούριο σε αυτό. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί περισσότερο είναι η διασύνδεση του στόχου τη νομισματικής σταθερότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μακροπρόθεσμα και τα δύο θα συγκλίνουν φυσικά. Διότι θα πει κανεί ότι αν έχουμε κανεί, για παράδειγμα τα πιστοτικά θέματα ακόμα και αν ο πληθωρισμό ε, ω επίπεδο είναι χαμηλός, όταν η φούσκα αυτή φουσκώσει θα υπάρχει μια νέα διάσταση όπου θα έχουμε ε, αν θέλετε μια νέα εξέλιξη ε, του ε, πληθωρισμού ίσως και με αρνητικές τιμές. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση μακροπρόθεσμα μεταξύ της νομισματικής σταθερότητας όπως την βλέπουμε με ένα σχετικά βραχυπρόθεσμο χρονορίζοντα και το θέμα της νομισματικής σταθερότητας. Το θέμα δημιουργείται όταν υπάρχει, όταν πρέπει να γίνουν επιλογές υπό συγκεκριμένε συνθήκες Μπορεί να έχει κανεί, ε, για παράδειγμα μέσα ε, των ε, ακινήτων ή των εξελίξεων στον πιστοτικό τομέα υπό εκρηκτική ανάπτυξη και βλέπουμε ότι σε σχέση όχι μόνο κοντοπρόθεσμα σε σχέση με την νομισματική σταθερότητα αλλά και μεσοπρόθεσμα σε ένα-δύο χρόνια υπάρχουν εξελίξει. Εκεί υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο στόχων καμιά φορά. Νομίζω ο σχεδιασμός των θεσμικών οργάνων που έχουμε σήμερα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που παραμένει στα πλαίσια της εντολής της, προσπαθώντας να κάνει καλύτερη χρήση του διπυλωνικού, της διπυλωνικής δομής, ε, διασφαλίζοντας και τα θέματα πιστώσεων. Αυτό προφανώς είναι μια δομή που πρέπει να διασφαλιστεί και να παραμείνει. Και όσον αφορά τις κεντρικές τράπεζες που εντάσσονται στον, στη διαχείριση του ευρωπαϊκού συστημικού κινδύνου, αποκινούμε τις άλλες θεσμικές αρχές. Γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου υπάρχουν νέες προκλήσεις και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της εντολή πρέπει να είναι σεβαστή. Δεδομένου το ότι παρεμβαίνει και στην νομισματική σταθερότητα η ΕΚΤ μαζί με άλλους ε, θεσμικά εμπλεκόμενου. Είναι κάτι που πρέπει από με πολύ προσοχή να εξετάσουμε. Έχουμε όμω το στόχο τη νομισματική σταθερότητα και τη αντιμετώπιση του πληθωρισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο ώστε αν χρειαστεί να ληφθεί δράση σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που ανέφερα στην εισαγωγή. Το σύμφωνο για το ευρώ. Μπορείτε να πείτε κάτι και για παρακαλώ. Ναι, για το σύμφωνο για το ευρώ. Νομίζω είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά πολλά πράγματα πιστεύω πρέπει ακόμα να αποσαφινιστούν στο τεχνικό, τεχνική υφή επίπεδο που πρέπει να διευκρινιστούν. Υπάρχει η γενική εντύπωση των κεντρικών τραπεζών ότι δηλαδή οι κανονισμοί, οι κανόνες δεν είναι αρκετά αυστηροί και στο σύμφωνο αυτό δεν υπάρχει επαρκής ε, αυτοματισμός ε, στις ε, διεργασίες. Εδώ υποστηρίζω εγώ προσωπικά αυτή την άποψη, όμως θα ήθελα αμέσω εδώ να προσθέσω κάτι. Κανόνες με αυτοματισμό κυρώσεων μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν υπάρχει θετική υποστήριξη από τους πολίτες, από τους λαούς μας. Μπορεί κανείς πολύ γοργά να περάσει σε λαϊκίστικες αντιδράσεις φυσικά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερο αυτοματισμό για την επιβολή κυρώσεων σε σχέση με αυτό το μηχανισμό. Ταυτόχρονα όμω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αντανακλάται αυτό και θα ενστερνίζονται οι πολίτε αυτή την προσπάθεια και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση όπω είπα. Βέρνερ, oh, παρακαλώ. Εσείς επανειλημμένα αναφέρατε ότι από του πολίτε πρέπει να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο το συστατικό αυτό, συνταγματικό α το πω έτσι, στοιχείο είναι η ανεξαρτησία όμω για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώ θα μετρήσετε αυτή την αποδοχή από του πολίτε χωρί να διακυβευτεί η ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι δύο τμήματα τη απάντηση άρρηκτα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό σε σχέση με το πολιτικό σώμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξηγήσει σε εσά το Ευρωκοινοβούλιο γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνε. Για παράδειγμα όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική και τους προϋπολογισμούς. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς γίνονται αποδεκτά από τους πολίτες. Τους πολίτες που εσείς εκπροσωπείτε ως αιρετοί εκπροσωπεί τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Και γι' αυτό δεν θα έχει αυτό. Δεν πρέπει να έχει επίπτωση αρνητική στην ε, ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να επεξηγείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί είναι σημαντικό και γιατί εμένουμε και επιμένουμε στον αυτοματισμό επιβολής κυρώσεων σε σχέση με την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων του χρόνου και Ανάπτυξης. Ε, okay, uh, ε, Ευχαριστώ. Ο διοικητής της ΕΚΤΑ μας προετοιμάζει ψυχολογικά για αύξηση επιτοκίων ενώπιον του πληθωρισμού κυρίως στην αγορά πρώτων υλών. Όμως, ο πληθωρισμός οφείλεται στο κόστος και όχι σε νομισματικούς παράγοντες. Πιστεύετε ότι αν γίνει αυστηρότερη νομισματική πολιτική ε, δεδομένη τη συγκυρία ε, είναι η καλύτερη δυνατή πολιτική για να αντιμετωπίσουμε πληθωρισμό που οφείλεται στο κόστο. Μήπω ισχύει το αντίθετο. Μήπω ε, δεν επιτρέψει περαιτέρω ανάκαμψη, κυρίως σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο ε, και σε περίοδο δύο δημοσιονομικής ε, λιτότητας και περιστολής των μισθών, ε, ε, διότι είπε ο κύριος Τρισί ότι θα ήταν λάθος να αυξήσουμε τους μισθούς. Οπότε τι γίνεται, έχουμε τρία φρένα, έχουμε λιτότητα σε όλους τους τομείς, στα δημόσια οικονομικά, στους μισθούς, στις τράπεζες και διαμορφώνουμε μία πολιτική που είναι εξαιρετικά προκυκλική, ενώ δεν έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της η παραγωγή των πρώτων υλών. Όταν θα συζητηθεί ενδεχομένω το ενδεχόμενο αυστηροποίηση εισαγωγικά της πολιτική, πώ θα τοποθετηθείτε εσεί, θα, απάντηση. Θα ήθελα να σχολιάσω όχι το τελευταίο θέμα που θίξατε, αλλά τη γενικότερη προσέγγιση. Κοιτάξτε, αυξάνεται το κόστο, ε, γιατί ε, αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή ε, πρόκειται για ένα αρνητικό σοκ, έτσι ονομάζεται αυτό. Αυτή είναι η χειρότερη δυνατή ε, περίπτωση γιατί αυξάνονται οι τιμές όταν είναι αρνητική ε, η προσφορά και μειώνεται και η παραγωγικότητα. Όταν αντίθετα έχετε σοκ που οφείλεται στη ζήτηση αυξάνονται οι τιμές αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Μα και τα δύο ισχύουν εδώ. Μα έχουμε σοκ ως προς τη ζήτηση επίσης, όχι μόνο ως προς την προσφορά. δίκιο έχετε απάντηση και αυτό περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα. Τέλο πάντων, όταν έχετε ένα τέτοιο σοκ αρνητική προσφοράς είναι δυσχερής η κατάσταση και βρισκόμαστε ενώπιον ενό διλήμματο. Τώρα, πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτό το σενάριο, αν η κατάσταση ε, είναι πρόσκαιρη ή μόνιμη ε, και αν συνεπάγεται μείωση επίπεδου ε, ζωής των χωρών καταναλωτών. Βέβαια, αυτό είναι θετικό για τι χώρε παραγωγού των πρώτων υλών. Αυτό είναι πολύ θετικό για αυτέ τι χώρε, αλλά το αντίθετο ισχύει για τι χώρε που καταναλώνουν. Οπότε, όταν υποβαθμίζεται το επίπεδο ζωής, γιατί ε, αυτό περιγράψατε στην ερώτησή σας, ε, πρέπει να δούμε αν θα το δεχτεί, αν θα το υποστεί μάλλον ολόκληρη η χώρα, ολόκληρο ο πληθυσμό ή όχι. Και ε, ποιο είναι το θέμα μας, αν το σοκ, οι δευτερεύουσες επιπτώσεις θα επηρεάσουν τις τιμές την πορεία των τιμών. Το πρώτο πρέπει να διαπιστώσουμε λοιπόν αν είναι πρόσκαιρη η κατάσταση ε, και στη συνέχεια να δούμε τη ροή των τιμών, το price flow. Ε, ναι, ποιες προσδοκίες υπάρχουν ως προς τον πληθωρισμό και ε, να υπολογίσουμε συνολικά το κόστος, όχι μόνο σε σχέση με τις τιμές, αλλά το συνολικότερο κόστος για την εθνική οικονομία λόγω της κατάστασης κατόπιν μπορώ να αμφισβητήσω αυτή τη διάγνωση που κάνατε σε σχέση με το ποσοστό χρήσης των παραγωγικών ικανοτήτων, του παραγωγικού δυναμικού. Ε, ε, ε, δεν Υπάρχει χαμηλό επίπεδο χρήσης ορισμένες φορές των παραγωγικών ικανοτήτων και να σας πω ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Ε, ε, εξαρτάται από τις χώρες. Κάποιες μεγάλες χώρες και κάποιες μικρότερες χώρες όπως η δική μου θεωρούν ότι σε αυτό το στάδιο του οικονομικού κύκλου χρησιμοποιούμε σε ικανοποιητικό βαθμό το παραγωγικό δυναμικό μας. Δείτε τις μεγάλες χώρες όπως ε, η Γερμανία ή μικρότερες χώρες όπως το Βέλγιο ε, να δείτε ότι το περιθώριο ελιγμών που έχουμε δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φανταζόμασταν. Ε. Το τελευταίο τώρα σημείο το ξέχασα. το ποσοστό χρήση του παραγωγικού δυναμικού. Δεν νομίζω να είπατε κάτι άλλο. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποια ερώτηση. Α, όταν έχετε ένα σοκ ανητικής ε, προσφοράς, ε, πρέπει να αναρωτηθούμε αν γίνεται ε, δεκτό από όλου, αν μπορεί να απορροφηθεί, αν θα μετακυλιστεί μέσω των τιμών, παραδείγματος χάρη, και θα επηρέασει άλλους τομείς οικονομίας. Α, θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι είναι μάλλον παρατεταμένη η περίοδος των χαμηλών ονομαστικών ε, τιμών 0,1% ε, τόσο κοντά στο 0 και ορισμένες φορές ε, περνάμε στο αρνητικό για, σε σχέση με τους κινδύνους. Ε, και το καταλογίζουμε αυτό στι βιομηχανοποιημένε χώρε. της είπα παραδείγματο χάρη, ότι είναι πολύ χαμηλά τα επίπεδα. Εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα ότι είναι σύντομη η περίοδος, αλλά δημιουργείται πρόβλημα για μια παρατεταμένη περίοδο, διότι ε, ε, ψάχνουν τα χρήματα διεξόδου επενδυτικέ και φυσικά με, χαμηλό, με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Ε, σε αυτή την αναζήτηση υψηλότερων επιδόσεων δημιουργούνται περαιτέρω πιέσει στο οικονομικό σύστημα. Ε, οπότε ε, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για μια μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Επόμενη ερώτηση από τον Wolf Klintz και να σας ρωτήσω μπορώ να δώσω τον λόγο στον προηγούμενο από εσά μπροστά σας γιατί πρέπει να αποχωρήσει. Ναι, συμφωνείτε. Ο Βούλφο πρώτος η χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικέ, όπως και κεντρικές άλλε τράπεζες δεν ήταν μόνο αρμόδιε ε, για την νομισματική σταθερότητα αλλά έπρεπε να επομισθούν μερίδιο για την ε, σταθεροποίηση και την ε, σταθερότητα των δημοσιονομικών και αυτό σε στενό συντονισμό με κυβερνήσει. Σε αυτή την περίπτωση πολύ σαφώ καταδείχθηκε ότι η ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά ήταν περιορισμένη και γι' αυτό η ερώτησή μου θα συμφωνούσατε ότι αυτό θα πρέπει ρητά να αναφερθεί και να συμπεριληφθεί στην εντολή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι όχι μόνο είναι αρμόδια για την σταθερότητα του νομίσματος αλλά και για την δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερον, η Ελλάδα θα έχει συσσωρεύσει, συσσωρεύσει εφέτος ε, χρέος 150-155% και θα γνωρίζετε ε, Σαπίρ και Μπρόγκελ ε, ανέλησαν αυτό και κατέληξαν στο σενάριο το, το αισιόδοξο ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτό το χρέος. Θα είσαστε εσείς υπέρ ότι θα πρέπει να υπάρξει εδώ μια ριζοσπαστική τομή. Δηλαδή στην Ελλάδα μέχρι 100% θα πρέπει να μειωθούν τα χρέη με ένα κούρεμα με τον ένα ή άλλο τρόπο και μετά θα ξεκινήσει μια νέα κίνηση από μηδενικό επίπεδο. Δεν έχει νόημα εδώ να αυταπατώμαστε και να αγνοούμε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη δεύτερη ερώτηση. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω και θα δώσω την κλασική απάντηση που, έχετε σε αυτό το, που αναμένετε σε αυτό το φόρουμ, αλλά πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα. Πάρα πολλές προσπάθειες έγιναν και πρόσφατα τώρα και στην Ελλάδα και έχουν συζητηθεί όλα αυτά. Χρειάζεται χρόνος πιστεύω και αυτό δόθηκε πρόσφατα με την επιμήκυνση της ε, εξόφλησης ε, του χρέους. Ε, την επιμήκυνση. Το είδαμε και σε άλλες χώρες ότι υψηλό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ όπως και το Βέλιο για παράδειγμα στο παρελθόν κατάφεραν με πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία δεν είναι τόσο μη ρεαλιστικά όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Όμως έχετε δίκιο στο ένα θέμα. Το κύριο θέμα για την Ελλάδα θα είναι η ανάπτυξη σε κάποιο σημείο. Αν η ονομαστική ανάπτυξη, ποσοστό ανάπτυξη θα είναι αρκετή για να μπορέσει να πάψει να εξελίσσεται σπυροειδώς αυτό το χρέος της. Δίνουμε μια ευκαιρία γι' αυτό. Θα δώσουμε χρόνο, παρέχουμε χρόνο. Είναι το πρώτο μέρος τη απάντησής μου, δεύτερο μέρος της απάντησης. Το μεγάλο θέμα των εξωτερικών παραγόντων, της αναδιάρθρωσης δηλαδή του χρέους. Θα έλεγα και σας υποβάλλω αυτή την πρόταση, αυτή την σκέψη σε εσάς και πρέπει να την αναλύσετε. Πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν αφήσουμε τέτοια κρατικά χρέη να ε, αποτύχει η απόσβεσή τους από κάποιες χώρες. Γνωρίζω το τι ε, συζητείτε. Λένε πολλές φορές ότι οι αρνητικές επιπτώσεις ε, εξωτερήκευσης θα είναι περιορισμένες σε σχέση με το σχεδιαζόμενο σενάριο. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στο πρόγραμμα της Ελλάδας που είναι πραγματικά πολύ σκληρό να πετύχει αλλά και η χώρα πραγματικά καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες. Να δοθεί ευκαιρία λοιπόν στην Ελλάδα να τα καταφέρει. Να μην λέμε δεν θα υπάρξει ποτέ επιτυχία, πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους ούτως ή άλλως. Οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ επώδυνες για τη χώρα ακόμα και σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Δεν υπάρχει δωρεάν διαδρομή. Για το άλλο θέμα είναι ένα πραγματικά φλεκτό, ε, ε, ε, φλέγον θέμα, πραγματική πρόκληση. Είναι ένα πραγματικά κέριο ζήτημα αυτό. Νομίζω μπορούμε να συγκεράσουμε και στο νομισματικό πλαίσιο της ανάλυσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουμε διπυλα, διπυλωνική προσέγγιση. Αν δείτε αυτή την προσέγγιση και δείτε τα, ισολογισμού τους ισολογισμούς σε σχέση με τις ε, πιστώσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς. Αν δείτε για παράδειγμα την ε, παροχή, την, α, ε, παροχή χρήματος, την προσφορά χρήματος την περίοδο πριν από την χρηματοοικονομική κρίση είναι σαφέ ότι στο μέλλον τέτοιου είδου πληροφορίε πρέπει να χρησιμοποιούνται στο νομισματικό πλαίσιο. Αν πάτε ένα βήμα όμω παραπέρα, είπατε θα πρέπει να επανακαθοριστεί η εντολή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. απαντώ κάθετα. Όχι. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Όποιο ε, αντιμετωπίζει το θέμα τη νομισματική σταθερότητα και τη αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αντιμετωπίζει πολυδιάστατα θέματα. Έχουμε τα θέματα των ε, ε πιστώσεων, του ε, χρέου. Είναι πολιτικά φλέγοντα θέματα. Αν αναμειχθεί κανεί σε αυτό, στο θεσμικό πλαίσιο, με τον όρο καθορισμού μια εντολή, τότε οι ευθύνε θα είναι θολέ, δεν θα είναι σαφεί και δεν συμβουλεύω να γίνει μια τέτοια ανάμειξη στην εντολή. Στην εντολή που έχουμε υπάρχει ε, περιθώριο να υπομισθούν από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των θεμάτων τη νομισματική σταθερότητα. Αλλά αυτό δεν είναι η αποκλειστική συνολική εικόνα. Βλέποντα αυτό πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προ το μέλλον περισσότερο και όχι μόνο στο παρελθόν και να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα στοιχεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μα στο παρελθόν. Αυτά είναι τα μαθήματα που πρέπει να συναγάγουμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, επειδή έχουμε και δύο ερωτήματα επ' αυτού. Το γεγονό ότι χρειάζεται ω ε, υπεύθυνο τη Κεντρική Τράπεζα κάποιο να έχει πληροφορίε από του επόπτε, τι ε, αρχέ εποπτεία. Καμιά φορά είναι εύκολο αυτό, γιατί καμιά φορά οι κεντρικέ τράπεζε ω επόπτε τραπεζών μπορούν ε, να διαχέουν αυτέ τι πληροφορίε στι συζητήσει για την νομισματική πολιτική. Δεν συμβαίνει όμω αυτό με όλε τι κεντρικέ τράπεζε. Και δεν συμβαίνει αυτό και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν έχει εποπτικό ρόλο σε σχέση με, τις με τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά ιδρύματα κατανοήσουμε το ρόλο αυτών όλων των εμπλεκόμενων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε τον μηχανισμό μετάδοσης ε, transmission mechanism και αυτό είναι εκείνο το οποίο σχεδιάζουμε και πρέπει να γίνει αλλά είναι τεράστια η πρόκληση φυσικά. Thank you. Gay. Thank you, Chairman. And thank you for... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με διευκολύνετε, μου δίνετε το λόγο τώρα γιατί ήρθε ο Υπουργό Οικονομικών της χώρας μου και θα πάω να το συναντήσω. Οι μόνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ευθύνε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Ιρλανδοί φορολογούμενοι, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεισέφερε στη δημιουργία του προβλήματος, γιατί πράγματι δεν είχε ακολουθήσει, εν πάση κάποιες προειδοποιήσεις οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει ούτε οι Ευρωπαίοι επενδυτές ε, οι οποίοι έβαλαν τα χρήματά τους στα πιστοτικά Ιρλανδικά Ιδρύματα. Ο φορολογούμενος είναι αυτός που πληρώνει το λογαριασμό. Εμείς περάσαμε από μια σχέση ΑΕΠ και χρέους από 30% σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο 120%. Κάτω από τις συνθήκες αυτές λοιπόν θεωρώ ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο ένας υπουργός οικονομικός μιας μεγάλης χώρας η οποία έχει σαν λόγω των εσωτερικών δυσκολιών τα δύο τρίτα του ύψους του φόρου ε, που επιβάλλει η Ιρλανδία στις επιχειρήσεις της ε, να καταγγέλει την κατάσταση της Ιρλανδίας και να την εκβιάζει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει καμία μορφή αλληλεγγύης και συνεργασίας εδώ. Θα δεχθείτε λοιπόν ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να να κουβαλήσει κάποιο βάρος το οποίο δεν είναι σε θέση να το κουβαλήσει λοιπόν και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, δεν είναι μια προσπάθεια αναζήτησης από διοπομπέων τραγών. Καταλαβαίνω την κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα εδώ σαν κεντρικός τραπεζίτης περισσότερο. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω ιδιωτικά μαζί σας για την κατάσταση αυτή, αλλά σαν κεντρικός τραπεζίτης δεν παρακολούθησα ακριβώς αυτά τα οποία είπατε για την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως είπα πριν, οι κεντρικοί τραπεζίτες γενικότερα θα έπρεπε να εξετάσουν ε, τους ε, χρηματοπιστωτικούς κύκλους πολύ περισσότερο από ό,τι το έκαναν μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο η κοινότητα των κεντρικών τραπεζιτών το έμαθε καλά το συζητήσαμε αυτό, είδαμε τους επιχειρηματικούς κύκλους, τους βλέπαμε αυτούς, αλλά όχι γενικά το χρηματοπιστωτικό θέμα. Για το θέμα των ευθυνών, το εύχραστο, το εύθραυστο των τραπεζών στην Ιρλανδία δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει ε, στα πλαίσια ευθυνών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέμα του πληθωρισμού, ναι, λέει ο κ. Μίτσελ, κοιτάξτε. Αυτό είπα, έπρεπε να είχαμε κοιτάξει περισσότερο τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους Οι πληθωριστικές τάσεις ε, ήταν περιορισμένες στο παρελθόν σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι έχουν κάποιες ευθύνες για την κατάσταση τη σημερινή, αλλά βάλατε σε πολύ ψηλό επίπεδο την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Σχετικά με το βάρος. Ε, δέχεστε ε, ότι αν μια χώρα ζητηθεί να αναλάβει ευθύνες τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για την Ευρωζώνη. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο του βάρους που μπορεί να φέρει μια χώρα. Κατανοώ τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα σας βέβαια, αλλά ένας από τους παράγοντες, και τώρα εκ των υστέρων είναι εύκολο να τα λέει κανείς, αλλά κάποιοι συνάδελφοι από τις κεντρικές τράπεζες και τις αρχές εποπτείας εργάζονταν για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης σαν και αυτήν την οποία περιγράφεται. Πώς μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που θα οδηγούσε στην μη δημιουργία των καταστάσεων αυτών θυμίζω ότι πριν από την κρίση είχαμε αφήσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα να αναπτυχθεί εντελώς ελεύθερα χωρίς τους μηχανισμούς επίλυσης των προβλημάτων. Και στα πλαίσια της Βασιλείας, του οργανισμού της Βασιλείας προσπαθήσαμε να δούμε τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί σήμερα και πολλές από τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο. Είναι μια τραγωδία αυτό το οποίο έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα κάνω την ερώτηση του συναδέλφου γιατί έπρεπε να πάει σε μια άλλη επιτροπή να παρουσιάσει την έκθεση. Λοιπόν, ε, η ΕΚΤΕ έχει το μεγαλύτερο κομμάτι δημοσίου χρέου σε διάφορα κράτη-μέλη και θα ήθελε να μάθει λοιπόν και θα διαβάσω την απάντησή σας ε, σχετικά με το τωρινό και μελλοντικό ρόλο των ε, CDS, ε, των μελλοντικών ασφαλίστρων κινδύνου. Ε, δύο ερωτήσεις ουσιαστικά θέσατε. Σχετικά με την πρώτη, η έκθεση η μόχλευση σε χώρες που αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες είναι μεγάλη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μην ξεχνάτε ότι ε, το μεγαλύτερο κομμάτι σχετίζεται με το double default, δηλαδή τη διπλή στάση πληρωμών. Όπως είδαμε και στη ΣΥΠΑ, ε, για να δοθεί ρευστότητα χρειάζεται εγγύηση, άρα χρειάζεται αυτό το double default για το μεγαλύτερο ε, τμήμα των κινητών ε, αξιών σας, το οποίο δεν ισχύει σε άλλα κομμάτια της αγοράς. Το δεύτερο ερώτημα τώρα που θέσατε για τα CDS Ε, άκουσα μία ερώτηση από τους πράσινους για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αν δείτε την γραπτή απάντηση που έδωσα, μίλησα για τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά. Ε, η αγορά των CDS εντάσσεται σε αυτό το μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν λειτουργεί ορθά ο μηχανισμός στην πράξη. Μπορείτε να αμφισβητήσετε τους τρόπους προσδιορισμού των τιμών. Πάντως εγώ σε, αυτόν τον γενικότερο, σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο εντάσσω το θέμα ε, των ασφαλίστρων κινδύνου. Πάντως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα ε, επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, επίσης για τις έξω συναλλαγές προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων για το συμψηφισμό. Του, τα CCPs δηλαδή. Ε, στα τέλη του 2012 ε, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ λεπτά ζητήματα. Έχουμε χρόνο, έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας, αλλά θα είναι εντατικέ οι εργασίες. Ε, πάντως για τα ασφάλιστρα Γνωρίζω ότι ε, το Κοινοβούλιο θέλει τις ε, ε, ακάλυπτες ανοιχτές πωλήσει να τις απαγορεύσει για τα CDS. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να καταργήσουμε τα naked ναι short selling, αυτές τις ακάλυπτες ανοιχτές πωλήσει. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένας από τους πράσινους. Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Ευχαριστώ, κύριε Πράιτ. Ευχαριστώ και για την απάντησή σα πριν. Μου δίνετε την αφορμή να σα ρωτήσω το εξή, Είναι γεγονός ότι χρειάζεται ανάπτυξη για την αποκλιμάκωση του χρέου. Όμω τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα δημοσιονομική προσαρμογή οδηγούν σε βαθιά ύφεση και αυτό δεν επιτρέπει δημιουργία πλεονασμάτων για να αντιμετωπιστεί το χρέο. Όμως ε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα, μια ανάγκη αποκλιμάκωση του χρέου, κυρίω για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. Οπότε θέλω να σα ρωτήσω Πώς ε, βλέπετε αυτή την ιδέα που συζητεί το Εβραίος πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν υπήρχε απόφαση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό, να δοθεί δυνατότητα στο μόνιμο ε, μηχανισμό σταθερότητας ή και στο προσωρινό ταμείο χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης να αγοράζει ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά να κάνει δηλαδή αυτό που κάνει σήμερα η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρευστότητας και ενδεχομένως να μπορεί να χορηγεί ε, το δάνεια στις χώρες για να επαναγοράζουν το χρέος τους. σας φαίνεται ότι αυτό είναι μια ιδέα που θα πρέπει να εξεταστεί μεσοπρόθεσμα; δεν εμπλέκομαι άμεσα στις τελευταίες συζητήσεις που έχουν γίνει για το ελληνικό χρέος. Αν κατάλαβα καλά τις ανακοινώσεις ορισμένων συναδέλφων μου από τις κεντρικές τράπεζες, θα πρέπει να υπάρξει ο μηχανισμός σταθερότητας, ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ ευέλικτος, να έχει ευρύτερη ευελιξία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Θα πρέπει όμως να κάνουμε εδώ μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα ταμείο το οποίο αγοράζει από τις αγορές απευθείας και να δανείζουμε ε, μια άλλη χώρα για να το κάνει η ίδια. Εγώ θα προτιμούσα τη δεύτερη μέθοδο λέγοντας ότι είναι καλύτερα να, αν χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό αυτό, να δανείσουμε μια χώρα έτσι ώστε να αγοράσει το χρέος της και μετά θα δούμε κατά από ποιες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο έκθεσης θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά αυτές οι επαναγορές τις οποίες βλέπετε συχνά στις ιδιωτικές αγορές είναι κάτι το οποίο αφορά αυστηρά την ιδιωτική αγορά. Όταν σε κάποιες εταιρείες έχουν προβλήματα με τράπεζες υπάρχει δυνατότητα επαναγοράς. Το ότι δηλαδή κάποιοι υποπίεση πολιτές θέλουν στη συγκεκριμένη περίπτωση να απαλλαγούν αυτό μπορεί να γίνει ε, βλέποντας όμως πρώτα τι τιμή ε, δίνει ο αγοραστής. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η αγορά θα αντιδράσει. Υπάρχει δυνατότητα. Ή μήπω η δυνατότητα αυτή είναι πάρα πολύ ακριβή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς την αξιολόγηση. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα έκθεσης ε, των ταμείων αυτών, διότι είναι δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα, δεν είναι πάντα διαθέσιμα οι συζητήσει, όπως είπα συνεχίζονται, δεν έχουν ολοκληρωθεί και στις οποίες συζητήσει θυμίζω ότι δεν συμμετέχω άμεσα. Θα πρέπει όμως να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιος μηχανισμός. Ο μηχανισμός σταθερότητας έχει αυτή τη στιγμή κάποια μέσα στη διάθεσή του ή τουλάχιστον αυτό έχει κυκλοφορήσει ε, στα μέσα ενημέρωσης. Όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πράτε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία, τη μία εύκολα θα την απαντήσετε, μονολεκτικά μάλλον. Ναι ή όχι. Όπως ε, Νόμιζα ότι η συνάδελφος Ιάννη Ποδηματά θα είχε κάνει την ερώτηση. Διάβασα τις απαντήσεις σας ε, και θεωρώ ότι πρέπει να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι ήταν σοφή η απόφαση του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα όταν ζητήθηκε η θέσπιση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θεωρείτε ότι ε, σωστά, σοφά αποφασίσαμε. Ε, απάντηση. Δεν είμαι μονολεκτικός εγώ στο ναι. στυλ μου. Μ' αρέσει να μακρηγορώ. Θα σας πω τα εξής. Δεν είμαι πεπισμένο ότι είχατε δίκιο. Δεν θέλω να κρίνω ούτε εσά ούτε το Κοινοβούλιο και τι αποφάσει που παίρνει, αλλά ακόμη δεν είμαι πεπισμένο για την ορθότητα του εγχειρήματο. Αλλά ε, ε, διαβάζοντας έγγραφα που εκπώνησε η Επιτροπή σα. Ε, τα βρήκα ενδιαφέροντα. Δεν είμαι πεπισμένο, το λέω, αλλά ε, υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Ε, και αν κατάλαβα καλά, θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί, να απαντήσει το κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή αυτού του μέτρου. Εμένα δεν με απασχολούν τόσο πολλοί φόροι, δεν είναι το δική μου αρμοδιότητα. εγώ όμω πρέπει να μεριμνήσω τόσο ώστε να μειωθεί η αστάθεια στι τιμέ και πώ θα αποφύγουμε με αυτό το φόρο την υπερβολική αύξηση των ε, τιμών ε, των κινητών αξιών. Ε, αν θα τα καταφέρουμε αυτά τα δύο μέσω του φόρου δεν είμαι επεπισμένος. Αλλά μπορούμε να το μελετήσουμε, να το διερευνήσουμε. Αυτή ήταν η εύκολη ερώτηση, κύριε Πρατείστη. Φιλελεύθερος μήπως και γι' αυτό έχετε μεσοβέζικη στάση. Δεδομένων των γεγονότων στην Ιαπωνία θα ήθελα να ε, ε, σχολιάσετε τις επιπτώσεις επί της νομισματικής πολιτικής, επί του πληθωρισμού και της εξέλιξης των επιτοκίων στην Ευρωζώνη λόγω των εξελίξεων. Γιατί αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε εσείς ε, την παρατήρησή μου. Μιλάμε για μια τραγωδία και νομίζω ότι τα πράγματα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπω κανείς τις τιμές στα χρηματιστήρια και τα λοιπά θα πρέπει ο καθένας από εμά σε προσωπικό επίπεδο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχει. Εμείς είχαμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις στην 11η Σεπτεμβρίου γιατί έπρεπε να παρέμβουμε άμεσα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρά την τραγωδία η οποία εξελισσόταν τότε. Ένα από τα πράγματα τα οποία είχαμε κάνει τις τελευταίες μέρες τότε ήταν να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υποδομές λειτουργούν σωστά στην Ιαπωνία. Μία από τις δικές μου ευθύνες, σαν παράδειγμα εδώ, όταν βλέπει κανείς ε, το σύστημα των συμψηφισμών με τις αντίστοιχες ε, Ιαπωνικές τράπεζες οι οποίες πολλούν ε, αξίες. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα πράγματα ε, συνεχίζουν και είμαστε σε επαφή με τις αρχές εποπτείας των υποδομών και με τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα συμψηφισμών στην Ιαπωνία τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και να σε ενημερώνουν σωστά. Για τις ευρύτερες επιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς. Ξέρουμε ότι το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που έρχεται στην επιφάνεια. Υπάρχει θέμα παροχής ενέργειας. Ξέρετε τις συζητήσεις που γίνονται και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες σε σχέση με την χρήση του πυρηνικού μέσου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται άμεσα στο νου. Ένα διαφορετικό θέμα αφορά κάποιες άλλες μορφές αβεβαιότητας. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλα προβλήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα στη διεθνή σκηνή η Μέση Ανατολή, οι επιπτώσει της χρηματοπιστωτική κρίσης. Έχουμε ένα επιπλέον επίπεδο εδώ θα έλεγα ανασφάλειας το οποίο συνήθως θα λειτουργεί αρνητικά για την ανάπτυξη. Αν συγκρίνει κανείς την κατάσταση με τον σεισμό του 95 δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να κάνει τη σύγκριση γιατί η κατάσταση δεν έχει ακόμα εξελιχθεί πλήρως δεν έχει ολοκληρωθεί θα έλεγα η καταστροφή. Αν δει κανείς το παρελθόν θα δει ότι η παραγωγή μειώνεται πάρα πολύ απότομα αλλά μετά αρχίζει και ανεβαίνει γιατί υπάρχει ανάγκη ανοικοδόμησης οπότε οι τιμές στα χρηματιστήρια, οι τιμές των μετοχών τουλάχιστον αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι για δύο μέρες έπεσαν πολύ και μετά αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν αυτό είναι το βασικό σενάριο αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι έχω τον τρόπο να αξιολογήσω τη σύνολη κατάσταση ένα άλλο θέμα είναι το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά όχι τώρα. Κοιτάξτε. Λίγο μεγαλύτερη πειθαρχία όσον αφορά τον χρόνο παρακαλώ τώρα. Επόμενη ερώτηση, εσύ, Γιώζεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία αποσαφήνιση. Αυτό το κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει μία πρόταση για τον μηχανισμό επίλυσης ε, τραπεζικών κρίσεων ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ρόλο του να συνεχιστεί η μερίσια διάταξη σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την κατάσταση σήμερα διατυπώνοντας μία ερώτηση να δούμε αν επιταχυνθεί το θέμα. Πρώτη ερώτηση. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την δυνατότητα, θα έχει εγκρίνει την δυνατότητα ο μηχανισμός για την αγορά του δημόσιου χρέους στον πρωτογενή τομέα. Θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αγοράζει κρατικό χρέος στις αγορές, στις δευτερογενείς αγορές ή θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει, να δίνει χρήμα στα κράτη-μέλη ώστε εκείνοι να εξαγοράσουν, εκείνα τα κράτη-μέλη να εξαγορέσουν το δικό τους κρατικό χρέος. η θα μπορουσε να συνεχισει να παρεχει να δινει χρημα στα κρατη μελη ωστε εκεινοι να εξαγορασουν εκεινα τα κρατη μελη να εξαγορεσουν το δικο τους κρατικο χρεος δεύτερη ερώτηση συγκεκριμένη. Η κοινή υποχρέωση σε σχέση με ένα όριο το οποίο δεν θα διακυβεύει τα δημοσιονομικά θα επέτρεπε να έχουμε μια αγορά πολύ μεγαλύτερη φερεγγιότητα, ρευστότητα όπω στην Αμερική, δίνοντα τη δυνατότητα να αυξηθεί η ζήτηση. Ποια θα ήταν η μείωση σε σχέση με το κόστος ε, της ε, ε, διαχείρισης, της έκδοσης, αν υπήρχε η δυνατότητα λειτουργίας μιας αγοράς αυτών των χαρακτηριστικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μου ζητήθηκε να είμαι και σύντομο στις απαντήσεις, δυστυχώς. Δύσκολη ερώτηση αυτή για το πρώτο. Σε σχέση με το μηχανισμό έχετε απόλυτα δίκιο. Σε όλη τη μεταρρύθμιση, τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση δεν προχωρήσαμε πάρα πολύ σε αυτή την πτυχή. Ακόμα και αν λάβει κανείς υπόψη την βούληση οι τράπεζες να μπορούν με μεγαλύτερη ας το πω ελευθερία να δρουν. Δεν έγιναν πολλά. Και μόλις ξεκινάμε σε σχέση με αυτό το στόχο, αυτό πρέπει να είναι μια κύρια προτεραιότητα. 100% συμφωνώ μαζί σας. Έκανε πολύ καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανε πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν υπάρχει μεγάλη όρεξη ως κίνητρο να προχωρήσουν όλοι. Και αυτό είναι πληρώνουμε το αντίτιμο του να είμαστε απροετοίμαστοι σε σχέση με αυτή την κρίση και δεν είμαστε ακόμα 100% σε θέση να συμφωνήσουμε ε, επ' αυτών. Αυτό είναι όμως μια κύρια προτεραιότητα. Δεύτερον, για το θέμα του αν θα πρέπει να δανείζονται, να υπάρχουν δάνεια, πιστώσεις για να αγοράσετε το ε, χρέος, το κρατικό χρέος. Σίγουρα θα πρέπει, διακόπτει ο μιλητής, παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται, εκτός μικροφώνου. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο πρωτογενή μηχανισμό θα λειτουργούσε, πώ και με ποιου όρου και προποθέσει. Είναι απόλυτα ασαφέ για μένα να απαντήσω σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σχεδιασμένη να αγοράζει στο δευτερογενή ε, τομέα, στο δευτερογενέ επίπεδο, εκτό αν μόνο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και για έκτακτη δράση μπορεί να εξεταστεί αυτό. Γι' αυτό έχουμε όλε αυτέ τι συζητήσει ε, και από ό,τι γίνεται αντιληπτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το τρίτο για το ευρωομόλογο και πάλι το ίδιο εδώ συμβαίνει και ως θέμα αρχής έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα είχαμε μια πιο ε, ε, μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά. Τώρα σε πώς, ε, υπάρχουν κάποιες αγορές που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα ή κάποιες άλλες που μπορεί να είναι ακόμα πιο υψηλά. Γιατί εδώ έχουμε και το θέμα, για παράδειγμα, του να δούμε την επίπτωση, την, τη διαμόρφωση των επιτοκίων που στη Γερμανία είναι χαμηλά, για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς πολύ αν δεν υπάρχουν τα αναγκαία κίνητρα. Ε, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα έκφραση τη αλληλεγγύη. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται εν ρευστό και γενικόλογα, χωρί ένα ισχυρό γενικό πλαίσιο που δεν υπάρχει σήμερα όσον αφορά κίνητρα. Γιατί αυτό είναι και η λίθο για την ε, ε, αλληλεγγύη. Ξέρω όλη τη συζήτηση για του διάφορου τύπου τύπους ομολόγων, αλλά οι όροι και οι προποθέσει είναι πολύ σημαντικά θέματα και δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συζητήσει επ' αυτών. Πρέπει να περιμένουμε να οριμάσουν. Η χρονική περίοδο δεν είναι ε, η πιο ευνοϊκή, δεν έχουμε τι απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Δύο ερωτήσει έχουν ε, απομείνει, Ελίσα και Άστριντ. Η Ελίσα πρώτη, παρακαλώ. σα ευχαριστώ πολύ. Πάντα είναι χαρά να ε, σα έχουμε ανάμεσά μα και η δική μου ερώτηση είναι η εξή. Για μας εκπροσώπου των Ευρωπαίων πολιτών είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια απάντηση όταν μας ρωτάνε οι πολίτες μας πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ανοιχτά την χρεοκοπία ολόκληρων χωρών της χώρας της ζώνης ευρώ όταν η Ευρώπη δεν ήταν ακόμα σε θέση να έχει μια δομή στη διάθεσή της επίλυσης των προβλημάτων, των τραπεζικών προβλημάτων, μεγάλων τραπεζών και υπερβολικά μεγάλων τραπεζών για τις χώρες όπου έχουν την έδρα τους. Και γι' αυτό, γι' αυτό το ερώτημα θα ήθελα, πέρα από το σχόλιο το οποίο κάνατε, να σας ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω για τον συνάδελφο κιόλας ε, Γκαρσία Μαργάλιο, να επεκταθείτε λίγο περισσότερο, μας πείτε κάτι παραπάνω. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν και σε σχέση με τη θέση σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι μπορεί να συνεισφέρει αυτό. Διότι έχουμε εδώ και το συστημικό κίνδυνο και εδώ πρέπει πολλή δουλειά να γίνει να αντιμετωπιστεί αυτό και βλέπουμε κάποιε κινήσει να γίνονται που δημιουργούν αρκετέ αμφιβολίες. Εμεί αγωνιζόμαστε και ε, εποφελούμεθα των γνώσεών σα ω πραγματογνωμονο για τα όσα έχουν προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια ευρωπαϊκή λύση δηλαδή, ε, banking, ε, European Banking Crisis Resolution, ευρωπαϊκή επίλυση τη τραπεζική κρίση και μέχρι στιγμή ε, η απάντηση βασίζεται σε μια ολόκληρη σειρά δημιουργία εθνικών ταμείων και όχι ενό Ευρωπαϊκού Ταμείου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αντίθετο δηλαδή αυτού που είχαμε εμεί προβλέψει και προτείναμε και σε σχέση με τι αποφάσει, τη προηγούμενη ενδεκάτη του μήνα βλέπουμε και εδώ άμεσα θα αναφερθώ στο ψήφισμα σε σχέση με τα συμπεράσματα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τη ζώνη ευρώ που λέει όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συγκεκριμένα προγράμματα θα συνάδουν με τους κανονισμούς και θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν με οποιαδήποτε τράπεζα θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, προβλήματα. Δηλαδή θα πρέπει αυτό σε σχέση με τα κράτη-μέλη να γίνει. Και συνεχίζει το κείμενο και λέει στην ενίσχυση της νομισματικής σταθερότητας θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να θεσμοθετήσουν εθνική νομοθεσία για την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου. Αυτό σημαίνει burden sharing, επιμερισμό βάρους και χρεών και εδώ είναι η ανάγλυφη ανάδειξη των επιπτώσεων αυτής της απαθίας που έδειξε η Ευρώπη. Well, uh, very much, uh, agree with, with, uh... Συμφωνώ, πολύ ε, με τις παρατηρήσεις σας επ' αυτών των σημείων και Απάντησα ήδη προηγούμενα μέρος αυτών. Δηλαδή δεν σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στο παρελθόν σε ένα κύριο θέμα το οποίο αφορά την ε, ε, αντιμετώπιση των θεμάτων της τραπεζικής κρίσης. Αυτό σύντομα επ' Το άλλο σημείο. Όταν θίγεται αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα, ακαθόδες θέμα, την εποπτεία της, ε, του χρηματοοικονομικού συστήματος, surveillance of the financial system, και μάλιστα εδώ θα ήθελα να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό έγκαιρα και σε, καλή, σε καλές ε, ε, συγκυρίες. Διότι όταν τα πράγματα οξύνονται, όπως και στο παρελθόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε να αποσταλούν ισχυρά αποτελεσματικά μηνύματα για φούσκες για παράδειγμα ή για ε, τα, τις τιμές ακινήτων κτλ. Όπως ξέρετε ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής Banking Supervision Committee στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όταν είχαμε το θέμα των, ε, ε, αυτών των φουσκών τότε εντοπίζοντας ε, σε μια χώρα το τι, ποια εξέλιξη σημειώταν, σημειωνόταν σε σχέση με τις τιμές, ε, ενώ οι εκπρόσωποι αυτής της χώρας έλεγαν «Α, δεν είναι τόσο αρνητική η κατάσταση, δεν γνωρίζετε ακριβώς τους, ε, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εξελίσσεται η αγορά μας». Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια αμερόληπτη, καλά πληροφορημένη πραγματογνώμονα αρχή, η οποία θα αποστέλει, θα δίνει αυτά τα μηνύματα έγκαιρα. Διότι όταν, έχει κανείς το θέμα των επιτόπου αρμοδίων, ακόμα και σε καλέ ε, περιόδους ε, είναι δύσκολο να αποσταλούν τα σωστά μηνύματα. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα αυτά στην πρακτική να λειτουργήσουν. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα πολιτική σημασία. Πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και αυτό είναι μία από τι μεγάλε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και το κατανοούμε απόλυτα αυτό. Το θέμα για την επίλυση τη τραπεζική κρίση που αναφέρατε και τι γίνεται με του πολίτε σε σχέση με αυτήν. Πολλά έχουν γίνει θα έλεγα. Αλλά τα κύρια ε, ζητήματα για την ε, ανθεκτικότητα του συστήματος ε, δεν έχουν επαρκώς απαντηθεί σήμερα. Έχουμε λοιπόν μεγάλη συζήτηση για τις απαιτήσει φερεγγιότητας και ρευστότητας, αλλά δεν έχουμε τόσα πολλά υποεξέλιξη για τον θεσμοθετημένο χαρακτήρα και σχεδιασμό των θεσμικών αυτών οργάνων και των ορίων τους. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε σε αυτό το πλαίσιο. Εκτό Εκτός από αυτά τα οποία συζητήσαμε πιο πριν για το CCP, για τις υποδομές έχουμε σημειώσει πρόοδος αλλά για τα άλλα θέματα δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Και για το πλαίσιο για την επίλυση των προβλημάτων έχετε απόλυτα δίκιο. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα πιο πριν. Δεν έχει συμμετεί πρόοδος. Αλλά δεν ρίχνω, ας πούμε, την εννοή. δεν ε, λέω ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είχε... έχει δραστηριοποιηθεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, συγγνώμη, δεν κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βλέπω ότι κινούμαστε από μια Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή λύση σε ένα σύνολο εθνικών λύσεων και αυτή η τάση είναι επικίνδυνη. Ο μιλητή συμφωνώ πολύ, διότι αναφέρατε την δυνατότητα ενό ευρωπαϊκού ταμείου που θα μπορεί να παρεμβαίνει σε σχέση με τα τραπεζικά αυτά θέματα. Ήμουν και στην άλλη αυτή η ομάδα εργασία Ευρωπα... στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Στην αρχή υπήρχε μεγάλη όρεξη λέγοντα, «Ε, ωραία, θα πρέπει να πληρώνουν οι τράπεζε ένα τέλο που θα πηγαίνει σε ένα τραπεζικό ταμείο για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Αυτό ήταν στην πρώτη φάση. Μετά αυτό εγκαταλείφθηκε. Αυτό σε σχέση με φορολογική ίσπραξη, α το πω, ε, τελών. Μετά έγινε εθνικού χαρακτήρα ότι ε, φορολογούνται επαρκώ οι τράπεζε, θα πρέπει να βρεθεί άλλο πλαίσιο δράση. Βλέπουμε ότι απαμβλήθηκε αυτή η όρεξη, αυτά τα κίνητρα σε σχέση με αυτή την ομάδα. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Τελευταία ερώτηση, η Άστριντ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τρισέ Μας είχε προειδοποιήσει κατά της εισαγωγής ενός φόρου στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Μας είχε πει επίσης εδώ και πολλές φορές μάλιστα καταδικάσει το σύστημα αυτόματης προσαρμογής των μισθών ε, στον δίκτυ του κόστου ζωής. Συμφωνείτε με τον κύριο Τρισέ σε σχέση με αυτό. Φυσικά, λέει ο κύριος Πανπράτ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ή για τον φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Θα πρέπει να ε, ερμηνευθεί. Αλλά σας είπα ποια είναι η όψη μου ή η άποψή μου ε, το πώς θα λειτουργήσουν τα επίπεδα των τιμών στις χρηματαγορές, οι υπερβολικές αυξήσεις τις οποίες βλέπουμε και το ότι κάποιες τιμές ξεπερνούν τη θεμελιακή τους αξία δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός τέτοιου φόρου συναλλαγών. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται στο Κοινοβούλιο είναι να βρεθεί μια συνταγή θα έλεγα και εμένα κάτι τέτοιο με ενδιαφέρει σαν κεντρικό τραπεζίτη. Εδώ θα έλεγα θα πρέπει να δούμε, να πω ότι η ποιότητα των, των στοιχείων που έχουμε έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα και η συζήτηση είναι πολύ πιο επαγγελματική από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια ας πούμε. Αξίζει λοιπόν, ίσως κάποιοι να το δοκιμάσουμε, αλλά είμαι σκεπτικιστής σε σχέση με τον στόχο που έχουμε, την λειτουργία των τιμών στις αγορές. Ο μηχανισμός αυτός κάλυψης των τιμών δηλαδή, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τον αφήσουμε να λειτουργήσει. Τώρα για την σύνδεση των μισθών με τον δίκτυ τιμών. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα στη δική μου χώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μην έχουμε κάποιο μηχανισμό είτε μηχανισμό διοικητικών σε εισαγωγικά τιμών, καθορισμού διοικητικού των τιμών, έτσι ώστε όταν υπάρχει ένα σοκ σαν παράδειγμα αρνητικής προσφοράς στις πρώτες ύλες να υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί. Και έτσι τα σοκ αυτά να προστατεύουν αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις αγορές, αυτοί οι οποίοι έχουν ας πούμε τις τιμές τους συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό σε σχέση με τους άλλους που δεν το έχουν. Νομίζω ότι ε, ένα τέτοιο σοκ αρνητικής προσφοράς είναι στην ουσία μια διαδικασία πτώχευσης της χώρας, πτώχευσης ενώ προοδευτικής, σταδιακής πτώχευσης και δημιουργείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό γιατί κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια σημαντική θέση περνούν την αρνητική αυτή προσφορά στους ε, συμβαλωμένους τους. Λοιπόν και στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο υπάρχει μια τέτοια μορφή σύνδεσης. Στο Λουξεμβούργο είχε προστατεύσει σαν παράδειγμα μετά το πρώτο πετρελαϊκό σοκ ένα τμήμα των εργαζομένων αλλά ένα άλλο τμήμα του παραγωγικού μηχανισμού υπέστη τις συνέπειες της αρνητικής προσφοράς. Στο Βέλγιο αλλάξαμε εμείς αυτόν τον μηχανισμό σύνδεσης για να μπορέσουμε να τον απομονώσουμε από τα σοκ αρνητικής προσφοράς βασική μου άποψη είναι ότι ο μηχανισμός σύνδεσης στο Βέλγιο δεν είναι αρκετά ισχυρός σε σχέση με τους μηχανισμούς αρνητικής προσφοράς. Και γίνεται μια συζήτηση στο Βέλγιο τώρα, έτσι ώστε να επανεξεταστεί αυτός ο μηχανισμός σύνδεσης, έτσι ώστε όταν υπάρχει μια τέτοια αύξηση στις πρώτες ύλε, ο μηχανισμός αυτός να μην περνάει πάρα πολύ γρήγορα το σόκο αυτό στο κόστος των επιχειρήσεων. Λοιπόν, όλα έχουν ε, σχέση με τις αρνητικές συνέπειες ενός σοκ. Όταν έρχεται ένα σοκ αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς και οδηγεί μέσω αυτής της σύνδεσης σε αύξηση των τιμών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα σαν παράδειγμα εξουδετέρωσης ε, κάποιων ε, τιμών στους δείκτες. Σαν παράδειγμα όταν αυξάνουμε τα τέλη για τον καπνό αυξάνεται ο πληθωρισμός. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να εξουδετερώσουμε κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε μέχρι τώρα υπόψη ή να καταργήσουμε το σύστημα αυτό. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν και ο μηχανισμός δεν εξουδετερώνει τις αρνητικές συνέπειες βλέπετε ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού στο Βέλγιο είναι υψηλότερος από τον μέσο ε, ρυθμό αύξησης της Ευρωζώνης. Υπάρχει όμως και το θέμα της ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς. Υπάρχουν οι λεγόμενες εισαγωγικά διοικούμενες ή καθοριζόμενες τιμές. Και επίσης οι πολύ ε, ικανές, ε, οι υψηλές θέσεις ορισμένων επιχειρηματικών εταίρων στις αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε μεμονωμένα και σε επίπεδο σύνδεσης των μισθών με το, κόστος, με το ύψος του πληθωρισμού, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις. Τέρμα. Θα έχουμε τώρα και κλεισμένων των θυρών μια συζήτηση μεταξύ ευρωβουλευτών. Εκείνοι που δεν είναι ευρωβουλευτές παρακαλώ να εγκαταλείψουν τώρα την αίθουσα. Εντάξει.